Ε, και πάλι, καλώς ήρθατε. Να καλωσορίσω τους αναφέροντες. Ε, χαίρομαι που είστε εδώ παρόντες. Και ελπίζω να έχετε υπομονή να μας ανεχτείτε, καθώς ε, θα πρέπει να συζητήσουμε ορισμένε διατυπώσεις εδώ στην Επιτροπή. Καταρχήν να περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση τη 11η Ιουλίου. Έχουν κυκλοφορήσει τα έγγραφα σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα. Μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Ωραία. Δεν ε, έχω ανακοινώσει στο σημείο αυτό. Ότι ε, ούτε έχουμε κάτι ποτέ διάφορα, όμως έχω πολλά να σας πω για τα αποτελέσματα της αποφάσεις των συντονιστών. Μία σειρά αναφορών θα προσθεθούν στην ουσία διάταξη του Νοεμβρίου, δεδομένου ότι έχουμε απάντηση της Κομισιόν. Και θα δείτε φυσικά όλα αυτά τα νούμερα τα είχαμε και στην ημερησία διάταξη των συντονιστών. Σε ό,τι αφορά το follow-up, στην ε, αναφορά για τα αγνοούμενα μωρά ή τα παχθέντα μωρά στην Ισπανία πριν πολλά χρόνια συμφωνήσαμε να καλέσουμε μία ή δύο οργανώσεις που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και να λάβουμε υπόψη και τη συνοριακή πτυχή. Θα έχουμε λοιπόν και κάποιον επιτρεμένο βασίλειο. Επίσης, συμφωνήσαμε να καλέσουμε την ε, Ombudsman, την Emily O'Reilly, στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου και συζητήσαμε και τις εργασίες της Επιτροπής για τους επόμενους μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία. Και τώρα προετοιμάσουμε ένα κατάλογο θεμάτων προτεραιότητας, ε, τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο και οι συντοριστές θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητές τους ε, πριν την προηγούμενη συνεδρία στις 8 Οκτωβρίου. Επίσης, ε, συμφωνήσαμε στην προτεραιότητα χρονοδιάγραμμα για την ετήσια έκθεση και την ετήσια έκθεση Ombudsman ε, του 2017. Αυτά να μπουν στην ημερησία διάταξη για την Ολομέλεια ήδη το Δεκέμβριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, συστάσεις, τις επίμαχες, υιοθετήθηκαν με την εξαίρεση της αναφοράς 0378 που θα παραμείνει ανοιχτή. Η αναφορά αυτή λοιπόν θα μείνει ανοιχτή και θα έχουμε follow-up για τα σημεία Β. Θα δώσουμε λεπτομέρειες γραπτός ε, για τις διερευνητικές αποστολές και κροάσεις. Ανταλλάξαμε απόψεις για το θέμα αυτό και θα λάβουμε μια απόφαση στην επόμενη συνεδρία του Οκτωβρίου. Επιπρόσθετα, οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι οι η διερευνητική αποστολή στην ε, Βαλεντόρα 17-18 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα και είμαστε ικανοποιημένοι να ανακοινώσουμε ότι ο συντονιστής ε, του ΕΛΚ, ο κύριος Γιάρ, θα συμμετέχει ο ίδιος και επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία. Συζητήσαμε την ε, κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με Συμβούλιο και Κομισιόν ε, για τον κανονισμό ECI και συμφωνήσαμε ότι ο για το άρθρο 14 που θα δικαταστεί στον κύριο Βαλέσσα είναι ο κύριο Πρέντερ από το ΕΛΚ. Η διάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων θα λάβει χώρα στις 27 Νοεμβρίου και σημειώσαμε ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα που έχει κυκλοφορήσει την περασμένη Πέμπτη. Επιπρόσθετα, η αναφορά 48 για την ατμοσφαιρική ρήπανση ε, στη Βαλένσια αποφασίσαμε να τη διατηρήσουμε ανοιχτή και να στείλουμε επιστολές στις Ισπανικές Αρχές. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συνεδρίασης των συντονιστών. Τώρα πάμε στο επόμενο σημείο που έχω εδώ να σας παρουσιάσω είναι να ψηφίσουμε ε, στην για την προφορική ερώτηση προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το ρόλο τη Γερμανική Υπηρεσία Πρόνοια Ανηλίκων. Να σας υπενθυμίσω ότι κατόπιν ετοίματος των σοσιαλιστών και του EFTD οι συντονιστές αποφάσισαν να καταρτήσουν ένα ψήφισμα ε, για το ρόλο της Jugendamt στη Γερμανία και λάβουν αυτή την απόφαση τον Ιούνιο. Τώρα το κείμενο είναι διαθέσιμο και καλούνται οι ομάδες ε, να καταθέσουν τροπολογίες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι συντονιστές έχουν λάβει απόφαση ότι το κείμενο θα είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά προκειμένου να προχωρήσουμε ταχύτερα με το θέμα αυτό. Αυτό επίσης σημαίνει ότι όλες οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά. Ελπίζω ότι θα συνεργαστείτε στενά προκειμένου να καταλήξετε σε συμβιβασμού. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ολομέλεια. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου και προτείνω προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Σημειώστε Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Έχετε λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί αρχικά, κατά δύο μέρες. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Και τώρα. Θα ήθελα να περάσουμε στην ψηφοφορία. What we actually are voting. Γεια σου, Ρομπέρτα. Ψηφίζουμε υπέρ ή κατά του κειμένου της προφορικής ερώτησης. Ποιος είναι υπέρ. S&D, πράσινη, EFTD. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Το ΕΛΚ απέχει. In favor of the text and as I... Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο. Όπως σας είπα, μπορείτε να το τροποποιήσετε όσο θέλετε. Η 28 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών, η επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Βιρζινή, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την προθεσμία. Μήπως θα ήταν δυνατόν η προθεσμία να πάει μέχρι την 1η Οκτωβρίου για τροπολογίες και με το at διοτι έχουμε να κάνουμε με ένα ψήφισμα που είναι σημαντική. Έχουμε 300 αναφορές. Πρόκειται για την εφαρμογή του δικαίου, το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών. Ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε εδώ και καιρό πρέπει να έχουμε όλες τις ευκαιρίες με το μέρος μας για να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα όσο γίνεται καλύτερο. Αναβολή της προθεσμίας για υποβολή τροπολογιών λοιπόν. Πρόεδρος, αν υπάρξει τέτοια αναβολή, ήδη έδωσα κάποιες μέρες. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερο χρόνο, αλλά τότε δεν θα πάει στην Ολομέλεια, τότε που είπαμε. Οπότε, ό,τι θέλετε αν θέλετε να αναβληθεί προθεσμία μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, αλλά τότε θα πάει στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Μα εγώ ήξερα ότι αν η προθεσμία πάει για την 1η Οκτωβρίου, μπορούμε να έχουμε το θέμα το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Μιλάμε για δύο μέρες παραπάνω, έτσι. Και αν γίνει με το 84M, τότε πιστεύω ότι Εφόσον δηλαδή στείλουμε online τι τροπολογίε, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το FDD ήθελε δύο μέρε. γιατί αρχικά ήταν 26 Σεπτεμβρίου. Και είπε το FDD ότι ήθελε δύο μέρε παραπάνω και είπε εντάξει. 28 Σεπτεμβρίου. Τώρα αν θέλετε παραπάνω, κάνει διαφορά, τι λέει η γραμματεία. Λοιπόν, έχουμε σχεδιάσει 9 Οκτωβρίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Αν βέβαια υπάρχουν πολλές τροπολογίες, δεν θα μπορέσει η γραμματεία να προετοιμαστεί μέχρι τότε. Οπότε μπορεί να πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, αλλά δεν είναι σίγουρο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ γεμάτη η Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Θα είναι δύσκολο για τη γραμματεία. Αν είναι λίγες οι έχει καλώς. Αλλά αν είναι πολλές οι θα είναι δύσκολο. Ωραία, αν είναι 28. Μπορούμε να υποβάλουμε τι τροπολογίες μέσω του συστήματος VTM, οπότε μπορούν να έχουν συνυπογραφεί ε, να μπορέσουμε έτσι να δουλέψουμε πιο εύκολα. Ιδίω αν κρατήσουμε την 28η Σεπτεμβρίου για να μπορέσουμε να πετύχουμε την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ωραία λέει η Πρόεδρος τότε. 1η Οκτωβρίου η προθεσμία. Στις 12 το μεσημέρι. Έτσι έχετε όλο το πρωινό Μα το βασικό μου αίτημα είναι να υπάρχει δυνατότητα μέσω του VAT4M να υποβληθούν οι τροπολογίε. Σε αυτή την περίπτωση ακόμα και 28 να είναι η προθεσμία, για μένα είναι εντάξει. Ναι. 1η Οκτωβρίου στις 3, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά μπορούμε τις τροπολογίες να τις υποβάλουμε μέσω του συστήματος online. 3 το μεσημέρι. Κυρία Πρόεδρε, δεν μιλάω για την ημέρα. Ρωτάω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής τροπολογιών. Αυτό ρωτάω. Η γραμματεία θα προσπαθήσει. Ωραία. Ψηφίσαμε ε, για την προφορική ερώτηση στην Επιτροπή. Συνεχίζουμε τώρα με το ψήφισμα για το ίδιο θέμα προς το Συμβούλιο αυτή τη φορά. Υπέρ, η ίδια πλειοψηφία φαντάζομαι κατά. Το ΕΛΚ. Αποχή. Ωραία. Η ίδια πλειοψηφία λοιπόν ε, όσον αφορά την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Ψηφίσαμε λοιπόν και όσον αφορά την ερώτηση προς την Επιτροπή και όσον αφορά την ερώτηση προς το Συμβούλιο. Καλώς. Το επόμενο θέμα είναι ε, το ψήφισμα. Μόλις ψηφίσαμε την προφορική ερώτηση, τώρα λοιπόν έχουμε εξέταση του ψηφίσματος, του σχεδίου ψηφίσματος. Αναρωτιέμαι αν θέλει κανείς να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι. Ελεονόρα. Grazie Presidente. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο για το σχέδιο ψηφίσματος ε, που καταρτίζει αυτή η Επιτροπή γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό το κείμενο θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθεί. Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε με εξαντλητικό τρόπο όλα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που ένα νέο σύστημα όπως είναι το γερμανικό ε, σε ό,τι αφορά το οικογενειακό δίκαιο και αναφέρομαι συγκεκριμένα ε, στο πώς λειτουργεί τον Γιούγεντα είναι ένα εντελώ επίμαχο ζήτημα και πρέπει να εμβαθύνουμε. Γιατί συνεχίζουν ε, να επιδεινώνονται τα προβλήματα που καταγγέλουν οι αναφέροντες και είναι πολύ άριθμοι μέσω των αναφορών στην Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο και κυρίως οι γονείς που δεν είναι γερμανικής υπηκότητας ε, έχουν αναφέρει πολύ σοβαρές διακρίσεις που έχουν υποστεί κατόπιν πρακτικών και διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει οι αρμόδιες γερμανικές αρχές. Και μεταξύ αυτών αναφέρουμε τον Γιγκεντάντ, έχουμε πάρα πολλές ε, οικογενειακές διαμάχες που έχουν σοβαρές συνέπειες ε, απέναντι σε ανήλικα παιδιά. Δεν ε, μπορούμε λοιπόν να θέτουμε σε κίνδυνο την ευμερία των ίδιων των παιδιών ούτε πρέπει να αμφισβητούμε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματο ε, χάρη, ε, το δίκαιο ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, το ε, δίκαιο στην προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πάνω από 10 χρόνια είχαμε πάρα πολλές έρευνες για το γερμανικό σύστημα και την υπηρεσία πρόνοια σε θέματα οικογενειακού δικαίου που έγιναν από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την δική μας Επιτροπή. Όμως ε, παρόλα, τις, ε, παρόλα τα αιτήματα που στείλαμε και στις γερμανικές αρχές και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο όλα αυτά έχουν μείνει νεκρό γράμμα και ε, βλέπουμε ότι ακόμα και οι συστάσεις που προέκυψαν από μια ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε εντός αυτής της Επιτροπής το Μάιο του 2017 εκπώνησε ένα λεπτομερές έγγραφο και περίχε μια σειρά συστάσεων, ούτε αυτές έχουν υλοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, παρόλο που υπήρχαν πολυάριθμες εκκλήσεις με το πέρασμα των χρόνων, απέναντι στις ε, γερμανικές ε, αρχές ε, βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση. Δεν ε, έχουμε διαθέσιμα στοιχεία, ούτε στατιστικά στοιχεία, συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τι πράγμα, συγκεκριμένα για την ε, έκβαση των δικαστικών ε, υποθέσεων ε, όταν είχαμε παραδείγματο χάρη το να ζητά την κυδαιμονία κάποιος και μιλάμε για περιπτώσεις όπου ένας γονέας δεν ήταν Γερμανός ή παραδείγματος χάρη ε, τις περιπτώσεις όπου ένας δικαστής δεν υιοθέτησε τις συστάσεις της Jugendamt. Έχουμε μία φορμαλιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο θέμα αυτό. Αρνείται δηλαδή το να προβεί σε μία ε, λεπτομερή ανάλυση για την κατάσταση αυτή. Αντιθέτως, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε το θέμα αυτό και γι' αυτό θα καταθέσουμε τροπολογίες επί του ψηφίσματος. Και θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σημαντικές τροπολογίες επί των οποίων πρέπει να εργαστούμε. Έχουμε ε, από ε, την πλευρά των γερμανικών αρχών, κάποια συμπεριφορά, δηλαδή έχουν σχεδόν ποινικοποιήσει τους μη γερμανούς γονείς. Βλέπουμε ότι έχουμε λυπή εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από άλλα κράτη-μέλη ε, και τις ευθύνες τους αναθέτουν κυρίως στον γερμανό γονέα και επίσης το ανήλικος ε, παραμένει σε γερμανικό έδαφος ε, ακόμη και σε περιπτώσεις ε, που έχουμε οικογενειακή βία ε, το χάρη, αν το παιδί πήγαινε στον άλλο γονέα, μόνο έτσι θα μπορούσε να αποφύγει τις πράξεις βίας. Έτσι λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι οι τροπολογίε που θα καταθέσω για αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ, η Βυρζινή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ουσιαστικές αναφορές που έχουν να κάνουν με το ίδιο ακριβώς θέμα. Έχουμε πάνω από 300 αναφορές για το θέμα και αυτό μας δίνει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα και τι αντίκτυπο έχει και σε επίπεδο δικαίου και σε επίπεδο ζώων. Γιατί εδώ έχουμε γονείς που στερούνται ε, τα παιδιά τους και το αντίστροφο. Ε, πάντοτε ένας χωρισμός είναι δύσκολος για όλους τους ενεχομένους, όμως αυτή η δυσκολία εδώ διπλασιάζεται γιατί έχουμε μία ε, δυσκολία στο πλαίσιο του δικαίου και της δικαιοσύνης γιατί ε, ουσιαστικά οι γερμανικές αρχές ε, πρόνοια ανηλίκο ουσιαστικά εισάγουν διακρίσει κατά των γονέων που δεν είναι Γερμανοί ή που δεν είναι κάτοικοι Γερμανία. Και Έχουμε πολλές αναφορές που ασχοληθήκαμε. Ε, οι γερμανικές αρχές δεν αναγνωρίζουν ε, τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με την κυδαιμονία των παιδιών. Θα θέλαμε να σταματήσει αυτή η προκτική προκειμένου ε, να υπερασπιστούμε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Έχουμε θετήσει και ένα ψήφισμα για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού σε πάρα πολλές ομάδες εργασίας εδώ και μήνες. Κι όμως

Πολύ λίγες ε, δράσεις ε, έγιναν για να διασφαλιστεί απλώς το ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 2 που ανήκει στο δικαιώμα. Είναι λοιπόν επιτακτικός όταν μιλάμε για διαζύγιο ζευγαριών διασυνερικών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κριτήρια υπόψη από τη δικαιοδοσία και θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα άρθρα 15 και 7 για να καθοριστεί ποια είναι η αρμόδια δικαιοδοσία ε, και για να μην αποκτά δικαιώματα δικαιοδοσία που δεν έχει. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ. Γι' αυτό ζητάμε με επιμονή και εδώ και πολλά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τι δικέ τη ευθύνες, να παίξει το ρόλο που τη αναλογεί, δηλαδή τον ορθό σεβασμό, τον σεβασμό του κανονισμού Βρυξέλλε 2. Εδώ και χρόνια η απάντηση που δίνει σε σχέση με τη δικαστική αρμοδιότητα των κρατών ε, μελών ε, μας δείχνει ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα εδώ γιατί η συνήθεια της απελπισίας είναι χειρότερη από την ίδια την απελπισία. Γι' αυτό εδώ το ψήφισμα θέλουμε να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά στην Κομισιόν το ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Ο ρόλος αυτός δεν μπορεί να χαίρει μιας επιφανειακής μεταχείρισης. Telephone is living its own life, obviously. Το τηλέφωνο έχει τη δική της ζωή, νομίζει, το συγγνώμη. Έχουμε και άλλους σκιώδεις, αλλά κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο. Να δώσω το λόγο λοιπόν στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, παρακαλώ. Or Mrs. Setti. I have... Ή την κυρία Σέτη. Έχω δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποφασίστε ποιος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, είμαι η Βαλέρια Σέτη, συντονίστρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει την Επιτροπή σα ε, για τη συνεχή τη προσήλωση πάνω στο θέμα αυτό και τι εργασίε τη για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Όσον αφορά τα τρία θέματα που απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο ψηφίσματος, ε, θα ε, Ζητάτε δηλαδή ε, πιο ακριβή ελέγχους ε, και συγκέντρωση δεδομένων. Θέλουμε να σας πούμε ότι το ουσιαστικό δίκαιο για τα δικαιώματα του παιδιού δεν εμπίπτει στο, ε, στο, στην, αρμοδιότητα αρμοδιότητες κομισιών, εμπίπτουν όμως στον κανονισμό Βρυξέλλες 2α και ε, σε άρθρο του κανονισμού αυτού προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα θέματα συγκέντρωσης δεδομένων ε, να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Όσον αφορά την έκκληση για περισσότερη κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, θα ήθελα να σας θυμίσω ε, το Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που οργανώνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου προσκαλούνται πάνω από 300 ενδιαφερόμενοι στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού και ο βασικός στόχος είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ε, ε, αλληλοδιδαχή κοινωνικών υπηρεσιών και αρχών προστασίας του παιδιού. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, συγκαλέσει ομάδα επιρογνωμόνων που έχει βασικό στόχο την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αλληλοδιδαχής. Ε, στην ομάδα αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων, τη ε, της λειτουργίας των εθνικών υπηρεσιών για ε, υπηρεσίες προ το παιδί. Επίσης, προωθείται η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, και σε διασυνοριακές υποθέσεις ε, σχετικά με την γονική μέρημνα. Παρέχεται κατάρτιση ή διευκόλυνση διμερών συναντήσεων μεταξύ κρατών μελών. Όσον αφορά το τελευταίο θέμα και την έκκληση για συγχρηματοδότηση και προώθηση πλατφόρμας που να παρέχει βοήθεια σε ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να ε, αυξήσουμε το δυναμικό ε, του δικαστικού τομέα και άλλων ε, επαγγελμάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας του παιδιού. Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δικαιοσύνη, μία από τις προτεραιότητες χρηματοδότησης είναι η βελτίωση της κατάστασης παιδιών ε, σε αστικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων μέσω καλύτερων διαδικασιών, ε, καλύτερης διεκπαιρέωσης των υποθέσεων ε, και καλύτερης εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου. Επίσης, έχει δοθεί χρηματοδότηση για διάφορα εργαλεία όσον αφορά τις διεθνείς απαγωγές παιδιών, τη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές οικογενειακές υποθέσεις και γενικότερα για την προστασία του παιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας, εάν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Α, Πέτερ, θέλεις να πάρεις το λόγο. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάποια επιχειρήματα. Υπόθηκε επανειλημμένα ότι το βασικό μας ε, ενδιαφέρον ε, είναι η ευημερία του παιδιού. Το ψήφισμα αυτό είναι ανεπαρκές και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι το παιδί ο αναφέρον. Ε, λέμε ότι μας ενδιαφέρει κυρίως το παιδί, αλλά δεν είναι το παιδί ο αναφέρον. Και θα αναφερθώ τώρα στο γερμανικό σύστημα όπου υποτίθεται ότι οι υπηρεσίες πρόνοιας ε, ανηλίκων στη Γερμανία ακριβώς σκοπό έχουν να διαφυλάξουν το συμφέρον του παιδιού. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου δύο γονείς αγωνίζονται και οι δύο για την ε, γονική μέρημνα. Έχουμε όμως ε, δύο πλευρές ε, επίμονες και κάποιος πρέπει να αποφασίσει ποιος θα έχει τη γονική μέρημνα. Πάντα ο ένας δεν, από τους δύο δεν είναι ικανοποιημένος. Αναπόφευκτο είναι και το εξή. Η διεθνή κοινότητα έχει ασχοληθεί με το θέμα. Έχουμε τη Σύμβαση της Χάγης. Και εφόσον θέλουμε να βρίσκεται στο επίκεντρο το παιδί, θα πρέπει αυτός που είναι πιο κοντά στο παιδί να έχει τη γονική μέρημνα, αλλά αυτό είναι προβληματικό σε περιπτώσεις όπου όχι μόνο τσακώνονται οι γονεί, χωρίζουν, αλλά πόσο μάλλον όταν μετακομίζουν ένας πολύ μακριά από τον άλλον. Εμένα πάντα με απασχολεί στι υποθέσει αυτές. Ότι δεν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς απέναντι στου αναφέροντε, δεν είμαστε δικαστήριο εμείς. Σε μια πολιετή διαδικασία δεν είναι σωστό να δίνουμε ελπίδες σε κάποιον γονιό τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την περίπτωσή του. Η Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ δεν είναι αρμόδια. σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ελεονόρα, you just had the Ελιονόρα, θέλεις τον λόγο? Ε, να ξέρεις ότι δεν έχουμε χρόνο, έτσι πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, αφού άκουσα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησα το λόγο. Και ξαναλέω, έχει την ίδια φορμαλιστική προσέγγιση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι σε ποια βάση οικοδομούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε όχι μόνο την ευημερία των παιδιών σε όλη την επικράτεια της Ένωσης γιατί εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που το αναφέρουν πολλοί άριθμοι αναφέροντες και αναφέρονται ακριβώς στο γερμανικό σύστημα του γερμανικού δικαίου αν δηλαδή δεν μπορούμε να προφυλάξουμε τις μελλοντικέ γενιές και τα παιδιά μας, τότε τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομούμε. Νομίζω ότι είναι μειοπική η προσέγγιση της Κομισιόν και δεν ε, λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συνθήκων και των αξιών αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Όσον αφορά αυτό το ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού, είχα την εντύπωση πως η ιδέα της πηξίδας είναι κάπως μονόπλευρη. Δεν είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με τα δικαστήρια, δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην κάθε οικογένεια ο αναφέρον ε, κάθε φορά συντάσσει την ε, αναφορά του και προφανώς και είναι μονομερής. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η άποψη της άλλης πλευράς ε, στο ζευγάρι, οπότε θεωρώ πως πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι δικαστικές αποφάσεις και πρέπει να ξέρουμε πού έχουν καταλήξει οι διαδικασίες, αν έχει υπάρξει έφεση, αν έχει φτάσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και η κατευθυντήρια γραμμή μας εδώ κάθε φορά είναι η δραματική τραγική περιγραφή της κατάστασης. Αλλά προσοχή, δεν πρέπει εμείς να αντιδράμε μόνο στη μία πλευρά. Πολύ συχνά οι άνθρωποι δραματοποιούν υπερβολικά την περίπτωσή τους και έχουν την τάση να παραβλέπουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μην τους βολεύουν. Δύσκολα θα κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι τόσο τυπική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί συναισθηματικά να αντιδράει. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάποιος ο οποίος υπερβάλλει στη δικιά του την περίπτωση, πώς να αντιδράσει κανείς αυτό. Όταν βλέπουμε λοιπόν τις διάφορες αναφορές που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα, ε, πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιες είναι οι διαδικασίες και ποιες είναι οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που γράφουν τις αναφορές αυτές ε, φοβούνται ότι θα χάσουν. Είναι ευάλωτοι. Οπότε περιγράφουν με δραματικούς όρους την περίπτωσή τους. Και συναισθηματικά και εμείς κινδυνεύουμε να αντιδράσουμε χωρίς να είμαστε αντικειμενικοί, χωρίς να έχουμε την αντικειμενική αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν όμως έτσι να αποφασίσουμε για την τύχη ενός παιδιού, βάσει δηλαδή συναισθηματικών κριτηρίων. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ κυρία Πετέρα. Ωραία, τότε να ολοκληρώσουμε ως εξή. Το ψήφισμα τώρα θα τεθεί στη διαδικασία τροπολογιών. 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, παρακαλώ, αυτά για την προθεσμία τροπολογιών. Και περνάμε στην επόμενη αναφορά, είναι η αναφορά 1018. Πρόκειται για μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων με πυρόληση στο πάρκο Πρασίνου του Στούροβο στη Σλοβακία. Έχουμε εδώ τους αναφέροντες, Στάμος Λεκοβίτς και Ντανιέλ Ζολτάι. Πού είσαστε? Που είναι οι αναφέροντες, παρακαλώ. Α, εσείς είσαστε. Ωραία. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Όχι ο καθένας, μαζί και οι δύο, έτσι. Ή ο ένας για πέντε λεπτά ή θα μοιραστείτε το χρόνο μεταξύ σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μα δώσατε να έρθουμε εδώ στη συνεδρίαση τη Επιτροπή σα, τώρα που συζητάτε την περίπτωση αυτή του Στούροβο στην Σλοβακία. Θα συνεχίσω στα σλοβακικά, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, ε, στα ουγγρικά θα συνεχίσω, λέει ο μιλητή. Είχαμε τρεις μέρες μόνο στη διάθεσή μας ε, στις, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκεντρώσαμε 8.000 υπογραφές για την περίπτωση του αποτεφρωτήρα αυτού. Και αυτό γιατί η τεχνολογία αυτή πυρόλησης ουσιαστικά ε, καίει απόβλητα. Δυστυχώς η μέθοδος αυτή δεν είναι πολύ καλή και θα επηρέσει αρνητικά ολόκληρη την περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρήπανσης. Ας δούμε τα γεγονότα. Η περιοχή αυτή είναι μια περιοχή με διάφορες ασθένειες. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή Υπάρχει ο Δούναβης, το Βίσεγκραφτ, ένα σωρό όμορφα μέρη και όμορφες πόλεις στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά υποφέρουν οι κάτοικοι από διάφορες ασθένειες. Εδώ βλέπετε μια πισίνα. Στην, ε, από τη Σλοβακία είμαστε περιοχή ε, που είναι η πιο ζεστή και υπάρχει δυνατότητα καλλιέργειας ε, αμπελιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να έχουμε μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ε, εδώ δίπλα. Είναι κάτι το οποίο θα χαλούσε όλη την περιοχή, θα κατέστρεφε όλη την περιοχή, η οποία βέβαια αποτελεί μεγάλη πηγή πλούτου για τον κόσμο που κατοικεί εκεί, τουρισμός, αμπέλια κλπ. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε τη βοήθειά σας. Αν έχουμε έναν από τα που δουλεύει εκεί, καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουμε. Θέλουμε να εμποδίσουμε λοιπόν αυτή την επένδυση, να μην υπάρξει μια τέτοια εγκατάσταση, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι πολύ αρνητικές στη ζωή μας. Εμείς θέλουμε να, ε, διατη... να προστατεύσουμε μάλλον τον μέλλον μας και να προσφέρουμε καθαρό αέρα στις μελλοντικές γενιές. Πολύ λογικά μου ακούγονται αυτά που λέτε. Θέλετε να διατηρήσετε τους σπόρους, ε, περιβαλλοντικές λοιπά για τις επόμενες γενιές. Πολύ καλό μου ακούγεται αυτό. Τώρα και εσείς, και εσείς θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που βάλατε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες και βλέπετε εδώ μια περιοχή με μνημεία, εθνικά μνημεία. Πρόκειται για έναν αγώνα που δίνουμε για την προστασία αυτού του εθνικού μνημείου στην πρώτη πρωτεύουσα της χώρας. Και όπως καταλαβαίνετε, το σοκ ήταν μεγάλο όταν ακούσαμε πως ένας τέτοιος αποτεφρωτήρας θα δημιουργηθεί στο Στούροβο και θα εγκατασταθεί στο Στούροβο. Αυτός ο αποτεφρωτήρας αποβλήτων από πλευράς τεχνολογίας έχει πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου, δεν υπάρχει τίποτα που να μας βοηθά να καταλάβουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην περιοχή. Αυτή η τεχνολογία πυρόλησης εξάλλου κάθε άλλο παρά η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία είναι για το σκοπό αυτό. Θα κάνει ζημιά στους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν η τοπική κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές παρενέβησαν στην διαδικασία εκ μέρους της Ουγγαρίας και το Υπουργείο Γεωργίας επίσης από όσο γνωρίζω έχει συγκεντρώσει πολλά έγγραφα. Θα ήθελα να θυμίσω, είμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν σε μια πόλη με τόσους ανθρώπους ουγγρικής καταγωγής να έχουν στην περιοχή τους ε, μια τέτοια εγκατάσταση χωρίς να έχουν ενημερωθεί. Όλα αυτά εμείς στοιχεία τα μάθαμε. Από όσο γνωρίζουμε, 17 θέσεις απασχόλησης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μόνο από αυτή την εγκατάσταση. Μόνο 17 θέσεις απασχόλησης. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο λοιπόν κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, θα μπορούσαμε και άλλες 8.000 υπογραφές να συγκεντρώσουμε. Οπότε σας παρακαλώ φροντίστε να σταματήσει ε, το σχέδιο αυτό για αυτήν την εγκατάσταση πυρόλησης και θέλω να σας πω ότι κάθε άλλο παρά μια καλή τεχνολογία είναι αυτή. Ευχαριστούμε. Τώρα. Μια στιγμή, γιατί έχω μπερδευτεί. Ναι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μίκελσον. Σωστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες ε, για τις εξηγήσεις που μας έδωσαν. Μπορώ να σας πω ότι το έργο αυτό εμπίπτει στην οδηγία για τις ε, ε, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη Μάλλον πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να υποβάλει απόψεις σχετικά με το έργο και όταν τελικά δοθεί η έγκριση από τις αρχές θα πρέπει να δηλωθεί πώς έχει ληφθεί υπόψη η κοινή γνώμη κατά τη λήψη της απόφασης. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που θέλω να πω. Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μόνο αφού ληφθεί απόφαση σχετικά με την οικοδομή και λειτουργία του έργου αυτού ε, μπορεί να γίνει κάτι μπορείτε νομίζω πιο αποτελεσματικά να παρέμβετε ε, με τις, τους μηχανισμούς που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Το έργο περιλαμβάνει αποτεφρωτήρα και ε, υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, εκπομπές ε, στον αέρα, το νερό, τα ύδατα και το έδαφος. Επιπλέον αναφερθήκατε στις βέλτιστες διαθέσιμες ε, τεχνικές και πράγματι υπάρχει η υποχρέωση να εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες. Ε, τι σημαίνει αυτό. Δεν μιλάμε για μία μόνο τεχνολογία μπορούμε, την οποία μπορούμε να επιβάλλουμε σε αυτούς που διαχειρίζονται την εγκατάσταση αλλά ε, τους υποχρεώνουμε να χρησιμοποιήσουμε να χρησιμοποιήσουν τις ε, βέλτιστες διαθέσιμε τεχνικές ε, για να ε, τηρήσουν το όριο των εκπομπών. Για τους τομείς που καλύπτει η οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει τεχνικούς κανόνες σχετικά με τις τεχνολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι εργασίες αυτές συνεχίζονται αυτή τη στιγμή και ένα πρώτο σχέδιο απόφασης θα συζητηθεί αρχές ε, του επόμενου έτους. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη διαδικασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να θέσει πιο αυστηρούς κανόνες για τέτοιου είδου εγκαταστάσει και τα σχετικά συμπεράσματα αναμένεται να υιοθετηθούν οριστικά τέλη του, έτους ή, ε, τέλη του επόμενου έτους ή αρχέ του 2020. Όπως σα είπα λοιπόν θα θεσπιστούν ακόμη πιο αυστηροί κανόνες ε, και ακόμα και οι διαχειριστές ε, υπαρχόντων μονάδων θα πρέπει να εφαρμόσουν του κανόνε αυτέ μέσα σε μια τετραετία. Ωστόσο, εάν δεν λειτουργεί ακόμη η εγκατάσταση που είναι το αντικείμενο της αναφοράς σας ε, κατά την υιοθέτηση των κανόνων αυτών, θα πρέπει ε, κατά την έναρξη λειτουργίας να συμμορφώνεται με τους κανόνες. Εάν λοιπόν ε, παρέμβετε την κατάλληλη στιγμή στη διαδικασία αυτή, θα μπορέσετε να διασφαλίσετε οι νέες αυτές εγκαταστάσεις ε, όχι μόνο να ε, συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή, αλλά και τους πιο αυστηρούς που θα τεθούν σε ισχύ στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Τσάκη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σλοβάκικα. Καταρχάς θα θέλαμε να επενέσουμε τις ενέργειες των αναφερόντων καθώς και την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πιστεύουμε ότι εκτιμάει πολύ σωστά την όλη κατάσταση. Αναφέρθηκε στις τεχνολογίες και εξήγησε πώς θα αξιολογούνται στο μέλλον οι τεχνολογίες αυτές. Έχοντας διαβάσει το υλικό και τα παρατήματα, Έχω εντοπίσει πέντε επίμαχα σημεία. Καταρχάς, ε, τεχνολογίες ε, και η μελλοντική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποτιμήσουμε την πτυχή αυτή. Άλλο θέμα είναι είναι η πιθανή κατάρρευση λόγω της ε, ισχύουσας ή της μελλοντικής νομοθεσίας. Τρίτον, έχουμε τον τουρισμό και το, τη διατήρηση του τοπίου είναι ένα ιδιαίτερα όμορφο τοπίο που επισκέπτονται τουρίστες από όλο τον κόσμο. Είναι ε, τοποθεσία με ε, έγκριση της UNESCO. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί. Επίσης βλέπω να υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στο ε, κοινό συμφέρον και τα συμφέροντα διαφόρων ομάδων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το κοινό συμφέρον και να του δώσουμε προτεραιότητα σε σχέση με τα συμφέροντα μικρότερων ομάδων, ε, ομάδων επενδυτών για παράδειγμα. Και τέλος, οι αναφέροντες ε, ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία ανάμεσα στις αρχές και στους πολίτες. ενδιαφέρον είναι ότι χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει την αναφορά αυτή και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πολίτες και των δύο χωρών έχουν υπογράψει την αναφορά. Τρεις προτάσεις έχω λοιπόν, Πρόεδρε. Να διαβιβάσουμε την ε, ε, αναφορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου μας και να ζητήσουμε τη γνωμοδότησή τους, να στείλουμε επιστολή στο Σλοβακικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ζητήσουμε τη δική τους θέση και τα σχέδια για το έργο αυτό. Και προτείνω επίσης να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την νομοθετική διαδικασία, όπως άλλωστε είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοψίζοντας λοιπόν, προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Μέχρι να διευκρινιστεί το θέμα. Ελπίζω να λάβουμε απαντήσεις από όλους τους σχετικούς φορείς αρχές του έτους και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην αναφορά αυτή έχοντας στα χέρια μας τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χελβένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου. Ως ε, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα και όχι στα συναισθήματα. Εγώ, ως ε, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, μπόρεσα να ενημερωθώ για αυτή την υπόθεση. Από ό,τι φαίνεται αυτή η επένδυση ε, θα ε, επεξεργάζεται 20.000 τόνους ε, προϊόντων στη μέση της πόλης. Και όταν η Κομισιόν αναφέρεται σε διάφορα σχέδια θα πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα της διαβούλευσης. Η διαβούλευση δεν έλαβε, δεν έλαβε χώρα. Θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα η διαβούλευση καταρχήν και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Όπως ε, είπα, ε, ουσιαστικά πρόκειται ε, για ένα εργοστάσιο, πρώην εργοστάσιο χάρτου, ε, και ε, πάρα πολλά χωριά και πόλεις ε, θα υφιστούν τις συνέπειες και από την πλευρά της Ουγγαρίας. Για να δούμε ξεκάθαρα, αυτό το εργοστάσιο θα χρησιμοποιήσει την πυρόληση ως μέθοδο και σύμφωνα με το Εθνικό και το Διεθνές Δίκαιο μιλάμε για έναν αποτεφρωτήρα αποβλήτων. Εδώ θα έχουμε οξύδια, ε, μονοξίδια και άλλα τοξικά υλικά που θα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Έχουμε ήδη κάποια εργοστάσια που λειτουργούν στην περιοχή και ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν και αυτό αποτελεί σορευτικό παράγοντα. Θα ήταν λοιπόν πολύ επιζήμιο στο περιβάλλον. Γι' αυτό αδυνατό να καταλάβω πώς ε, θα ήταν δυνατό να δοθεί έγκριση για μια τέτοια εγκατάσταση που θα χρησιμοποιεί την πυρόληση που θα έθετε ε, σε κίνδυνο την υγεία 40.000 κατοίκων στην περιοχή αλλά και ε, θα είχε και επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την αμπελοκαλλιέργεια. Μαζί με τον συνάδελφο, τον κύριο Τάκη, έχουμε υποβάλει μια γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν λάβαμε μία απάντηση που δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω τώρα εδώ, αλλά από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν δεν πιστεύει ότι είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Οι ντόπιοι διαμαρτυρήθηκαν και φυσικά μπορεί να προβλέψει κανείς ποιε θα είναι οι επικίνδυνε συνέπειες ε, μια ε, τέτοιας μονάδας. Η Κομισιόν όμως δεν άκουσε αυτή τη διαμαρτυρίες εδώ. Ε, μιλάμε για μια διασυνοριακή παράνοια. Πρέπει να ελέγξουμε πολύ σοβαρά τι γίνεται εδώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σα. Μπορείτε πάντοτε να εμπιστεύεστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι θα υπερασπίζουν το περιβάλλον, θα προστατεύουν το περιβάλλον όπω πάντα. Τώρα, α επανέλθουμε στου αναφέροντε. Όχι. Και ο Πίτερ θέλει το λόγο, παρακαλώ. Μία μικρή παρατήρηση. Είχαμε παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν και εμένα αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση είναι που οι αναφέροντες είπαν ότι κατά σύμπτωση ε, ενημερώθηκαν. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, αμοιβαία υποχρέωση πληροφόρησης. Σε περιπτώσεις όπου δημιουργούνται μονάδες στα σύνορα θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης. Η ε, υποχρέωση ενημέρωσης υπάρχει μόνο όταν έχουμε ε, προστατευόμενες περιοχές, προστατευόμενους οικότοπους. Η απόφαση δηλαδή παραμένει της ε, Σλοβακίας Θα πρέπει να ε, ε, ενημερώνεται η άλλη πλευρά. Σε άλλους τομείς πρέπει να ενημερώσω τον γειτονά μου για το τι κάνω στο σπίτι μου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερου κανόνε από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πολλά προβλήματα. Ε, καλώ την ε, Πρόεδρο να το λάβει αυτό υπόψη και να υπάρξει σχετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Διότι δεν είναι ικανοποιητικοί οι κανόνες που ισχύουν σε περιπτώσεις τέτοιων μονάδων, δημιουργήσατε τέτοιων μονάδων σε ε, ε, μεθόριες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώσαμε τους ομιλητές ε, στο θέμα αυτό και καλό τους αναφέροντες να ξαναπάρουν το λόγο και να απαντήσουν στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να σας απευθύνω μία έκκληση που είναι η εξής. Βάσει των επιχειρημάτων που ακούστηκαν, σας ζητάμε να ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό, γιατί ακόμη και αν αυτός ο δεν λειτουργεί ακόμη, ο επενδυτής κάνει τα πάντα προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του. Θέλουμε εμείς να σταματήσει αυτό το έργο και θέλουμε να αποφύγουμε όλες τις αρνητικές συνέπειες επί των ζώων μας και της υγείας μας. Θέλουμε να διατηρήσουμε την περιοχή μας καθαρή και έτσι να βοηθήσουμε και τις επόμενες γενιές. Επίσης, να αντιδράσω και εγώ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συνεισφορά σας. Και εγώ πιστεύω ότι είναι παράλογο να μην υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη νομοθεσία. Είμαστε κατά της ρήπανσης και της μόλυνσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και πολύ έξυπνα το έθεσε ο αναφέρον. Πρόκειται για ένα διασυνοριακό ζήτημα γιατί το νερό και ο αέρας δεν έχουν σύνορα. Έτσι λοιπόν είναι ένα πολύ καλό συμβολικό ζήτημα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό, να το επιλύσουμε σε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα. Και νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και πρότεινε ο συνάδελφο ότι θα πρέπει να προωθήσουμε στην ΕΝΒΗ για γνωμοδότηση ήδη. Του ενημερώσαμε. Μπορούμε να του πούμε ότι θέλουμε και εμεί να διερευνήσουμε το θέμα και να υπάρξει και μία γραπτή γνωμοδότηση στην Επιτροπή και να στείλουμε φυσικά και μία επιστολή στην κυβέρνηση της Σλοβακίας και να είμαστε σε στενή επικοινωνία με την Κομισιόν για το θέμα αυτό, γιατί η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακα των συνθήκων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς ανθρώπους. Επίσης, θα βάλω στην επιστολή τη σημασία των, ε, να γίνεται η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάτι που σέβεται τη Σύμβαση Άρους. Θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους θυγόμενους πολίτες, με τον κατάλληλο τρόπο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα λοιπόν που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε σε αυτή την επιστολή. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε. Συμφωνείτε όλοι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλή επιστροφή στη Σλοβακία και στην ωραία γωνιά της Ευρώπης. Συνεχίζουμε λοιπόν και ερχόμαστε στην ε, ερευνητική αποστολή που έλαβε χώρα στο Αθηνικό Δρυμό της Ντονιάνα πριν από λίγες μέρες. Ο κύριος Τσάκη ήταν επικεφαλής, οπότε θα σας δώσω και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στα Ουγγρικά. Όντως, περάσαμε τρεις μέρες στην Ισπανία και είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ την γραμματεία που οργάνωσε την επίσκεψη αυτή και ευχαριστώ πολύ και τους συμβούλους μας. Συναντηθήκαμε με τους αναφέροντες επιτόπου. Συναντήσαμε και εκπροσώπους των τοπικών οργανώσεων στη Σεβίλη. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, στον εθνικό αυτό δρυμό υπάρχουν κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα και υπάρχει κίνδυνος ρήπανσης του περιβάλλοντος και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι επίσης πολύ σοβαρό. Στην Ισπανία και κυρίως σε αυτή την περιοχή υπάρχει πρόβλημα έλλειψης υδάτινων πόρων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, όπως επίσης και η παράνομη χρήση των υδάτινων πόρων. Χρησιμοποιούνται δηλαδή παράνομα πηγάδια, φράτια και Φυσικά υπάρχει μεγάλη γεωργική δραστηριότητα. Όταν ε, χρησιμοποιούνται παράνομα ε, υδάτινοι πόροι, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι τις θερούνται άλλες περιοχές. Και ότι μπορεί να στερέψουν κάποια στιγμή οι πηγές αυτές. Οι αρχές λοιπόν και οι εκπρόσωποι της Ισπανικής κυβέρνησης είπαν ότι η παράνομη χρήση υδάτινων πόρων πρέπει να σταματήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ήδη έχουν κλείσει 350 φρεάτια και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η διαχείριση των υδάτων μπορεί να συνεχιστεί μόνο με συντεταγμένο τρόπο και νόμιμα. Ένα άλλο πρόβλημα, ίσως ακόμα πιο σοβαρό, είναι ότι πρόκειται για έναν εθνικό δρυμό, όπως είπα. γίνονται εξορίξεις στην περιοχή αυτή και οι περισσότεροι πόροι έχουν ήδη εξοριχθεί, παρόλα αυτά συνεχίζονται οι εξορίξεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και είναι πρόβλημα ε, βέβαια αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ε, γίνονται εισαγωγές από την Αφρική φυσικού αερίου σε αγωγούς υποπίεση δραστηριοποιούνται διάφορες εταιρείες και κάποια εταιρεία αποφάσισε ότι τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να αποθηκευτούν σε, παλιές, σε παλιούς χώρους δεξαμενές που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον φυσικό δρυμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι από σεισμού που γίνονται στην περιοχή αυτή μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Ένα τέταρτο πρόβλημα είναι οι αγροτικές δραστηριότητες. Έξω από αυτό το φυσικό δρυμό, και εδώ μιλάμε για ένα πολύ καλό έδαφος, πολύ καλή γη, υπάρχουν πολλές γεωργικές δραστηριότητες. Και όλες αυτές συνεχίζονται όχι μόνο εκτός του φυσικού δρυμού αλλά και μέσα. Και υπάρχουν μεγάλες απαιτήσει σε υδάτινους πόρους. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και με εξέπληξε θετικά θα έλεγα και όλους μας στην ε, αντιπροσωπεία που πήγε το γεγονός ότι οι οι τοπικές αρχές στην ε, Ανδαλουσία και στη Σεβίλη συμφωνούν. Δηλαδή βλέπουν το ζήτημα με τον ίδιο τρόπο. Υπήρξε πολιτική αλλαγή. Ο νέος υπουργός είναι ιδιαίτερα απόλυτος, δέχεται τα επιχειρήματά μας, οπότε οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά. Παραμείναμε στα γεγονότα. Έπειτα συναντηθήκαμε και με εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί λοιπόν μας εξήγησαν πώς διερευνούν τα διάφορα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα είναι η διαμάχη ανάμεσα στους γεωλόγους, τους εμπειρογνώμονες και τις ε, τοπικές ε, και εθνικές αρχές. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά στα δύο επίπεδα και μας είπαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας ε, σεισμός 3-3,5 ρίχτερ. Δηλαδή, οι γεωλόγοι τοπικοί είπαν ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Όμως οι εθνικοί γεωλόγοι λένε ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ακριβώς επειδή υπάρχει αποθήκευση φυσικού αερίου και μπορεί έτσι να υπάρξει διάβρωση και το αποτέλεσμα ε, αυτής της διάβρωσης μπορεί να είναι μεγάλο άπαξ και υπάρχει σεισμός. Επ' αυτού λοιπόν είναι που δεν συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες. Η εταιρεία λοιπόν διαθέτει 16 χώρους αποθήκευσης σε τέσσερα κομμάτια μοιρασμένα. Μία τέτοια αποθήκη, μικρή βέβαια, τηρεί τους κανόνες και έχει εγκριθεί από τις εθνικές αρχές. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όμως, οι τοπικές αρχές της Σεβίλη και οι κάτοικοι είναι κατά αυτών ε, των αποθηκών φυσικού αερίου. Είναι ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα, ιδιαίτερα επίμαχο. Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε τον ίδιο το Δρυμό, που είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη περιοχή. Ακόμα και αν τώρα είναι περίοδος ξηρασίας, δεν μπορέσαμε να τα δούμε όλα, ήταν ε, όμορφα. Και μετά πήγαμε στη Μαδρίτη και συναντήσαμε τις εθνικές αρχές. Ε, όπως σας είπα, υπήρξε πολιτική αλλαγή στην ε, Ισπανία και η νέα ισπανική κυβέρνηση τώρα δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, απάντησε στις ερωτήσεις μας, οπότε θα έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι ιδιαίτερα θετικό και με συστάσεις και ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε σύντομα. Οπότε ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή και πραγματικά είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Εσάς ευχαριστώ ε, που μας ε, περιγράψατε τα στοιχεία της επίσκεψης αυτής. Ε, ήταν δύσκολη η αποστολή. Ο κ. Μασελέης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ευχαριστώ τον Πρόεδρο της, επιστο... Αποστολής, ε, τόσο και για το έργο του κατά τη διάρκεια της Αποστολής και για τη σύνοψή του. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Καταρχήν ε, η συνεδρίαση με το νέο ε, Υπουργείο Περιβάλλοντο στην Ισπανία ήταν πολύ θετική, μας υποδέχτηκαν θετικά, αλλά ε, ακούσαμε και κάτι θεμελιώδες. Ήταν να δούμε ότι το σχέδιο αερίου στο πάρκο Ντονιάνα δεν είναι στρατηγικό σχέδιο για την Ισπανική κυβέρνηση. Ήταν στο παρελθόν, τώρα δεν είναι. Έτσι λοιπόν, ε, προκειμένου η Ισπανική κυβέρνηση να μπορέσει να ξεφορτωθεί το σχέδιο, το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ο εκφοβισμό που ασκεί η αρμόδια εταιρεία. Έτσι λοιπόν, εδώ μπορούμε να παίξουμε έναν θετικό ρόλο, να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση προ αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να βρει τρόπου ε, για να μπορέσει να ξεφορτωθεί ένα έργο που δεν είναι είναι στρατηγικό και μάλιστα βρίσκεται και κοντά στο Εθνικό Πάρκο και να βρει τρόπους ε, να μην ε, πληρώσει αποζημίωση γιατί τελικά ε, δεν πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες μέσω του λογαριασμού του ρεύματο. Επίση, μου φαίνεται πολύ σημαντικό ο ρόλο που παίζει το Κοινοβούλιο στο πρόβλημα του νερού. Κάθε φορά βλέπουμε ότι έχουμε πολύ σοβαρό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων γεωργία στην περίπτωση αυτή γύρω από τον Εθνικό Δρυμό με τα παράνομα ε, φρεάτια. Και πάλι εδώ οι αρχές ε, και από την τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας αλλά και από την κυβέρνηση είχαμε ε, μία δέσμευση για να τεθεί τέλος ε, σε αυτά τα φρεάτια. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία γιατί διαφορετικά, όπως μας είπαν στον Εθνικό Δρυμό, θα έχουμε πολύ σοβαρό αντίκτυπο για το ίδιο το Εθνικό Πάρκο αλλά και για τον περίγυρο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν ιδιαίτερα καρποφόρος αυτή η υποστολή. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κοινά ε, συμπεράσματα και η έκθεση που θα κάνουμε σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αναφέροντες αλλά και την τοπική αυτοδίκηση γιατί χρειάζεται αυτή η όθηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο πάνω στο θέμα αυτό. Άλλωστε, ο επικεφαλή τη αποστολή ε, μα περιέγραψε πολύ καλά το τι συνέβη και τι δεν συνέβη. Είχαμε επίση ε, μία επίσκεψη στην Λουσατία φέτο τον Φεβρουάριο, όπου επίση ήταν επικεφαλή ο κύριο Τσάκη. Θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε σύντομα. Όσο πιο σύντομος ε, μπορείτε να είστε, τόσο το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα είμαι σύντομος. Διότι Ήδη έχουμε συζητήσει δύο φορές το θέμα. Ε, εδώ ε, έχουμε χρήση άνθρακα για βιομηχανικούς σκοπούς και υπάρχει σύγκρουση με την τοπική κουλτούρα. Είναι κάτι το οποίο βλάπτει το περιβάλλον. Έχουμε εκπονήσει μια πολύ καλή έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία γι' αυτό. Είναι τόσο καλή η έκθεση που Ζητήσαμε παρατηρήσεις από τους Γερμανούς ε, συναδέρφους ε, και νομίζω ότι μόνο δύο παρατηρήσεις είχαν. Είναι λοιπόν έτοιμη η έκθεση, ισορροπημένη, είναι καλά καταρτισμένη και διαπεί επαγγελματικό πνεύμα. Στι 9 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές ελπίδες ότι θα υπερψηφιστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Στανόκα ε, συμμετείχε στην στην αποστολή αυτή. Δεν είναι πια ευρωβουλευτής, ε, είναι ε, στο, ε, στην πατρίδα της. Αλλά Μάργαρετ, θέλεις κάτι να πεις. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ, αλλά κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ αργά. Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε η αποστολή. Και νομίζω ότι οι άλλες εκθέσεις έχουν εκπονηθεί πολύ πιο σύντομα από αυτήν εδώ πέρα. Είναι πολύ αναλυτική η έκθεση και πολύ καλό το αποτέλεσμα. Απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι θα υποβάλω τροπολογίες, θα αναζητήσω συμβιβαστική λύση, αλλά σε ένα σημείο θα ήθελα να ε, έχουμε πιο ισχυρή διατύπωση. Εγώ συγκλονίστηκα που διαπίστωσα ότι δεν έχει αναλυφθεί καμία πρωτοβουλία να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ε, του μέλλοντος. Ε, συνεχίζεται η χρήση λιγνίτη. Και αν σκεφτούμε πόσοι μας μίλησαν ε, για το κοινωνικο-οικονομικό σοκ της Ανατολικής Γερμανίας, τι έγινε όταν κλείσαν όλοι αυτοί οι χώροι εργασίας, τι έγινε στην οικονομία. Εμένα με εκπλήσει το ότι τώρα ξεκινάνε να το σκέφτονται αυτό, αλλά ουσιαστικά τρεκλίζουν και θα φτάσουν σκοντάφτοντα σε μια παρόμοια κατάσταση. Είδαμε τον αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Φυσικά είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο κόσμο στην περιοχή αυτή, αντί απλά να περιμένει το μέλλον, να επενδύει ένα σωρό κεφάλαια σε βελτίωση των παλιών τεχνολογιών ε, της χρήσης ε, λιγνίτη που είναι ουσιαστικά το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. Ήθελα λοιπόν απλά να σας προειδοποιήσω ότι θα προσπαθήσω να καταρτήσω μια τροπολογία και ελπίζω να την στήριξει η Επιτροπή μας. Διότι νομίζω έχουμε και κάποιο είδους ευθύνη απέναντι στους πολίτες του μέλλοντος και όχι μόνο να κοιτάμε το βόλεμα όσων βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την τροπολογή υπολογιών στα αγγλικά μόνο θα είναι 26 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα το απόγευμα. Αυτή την Τετάρτη δηλαδή, ε. Και ψηφοφορία στις 9 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το σχέδιο έκθεσης και τις συστάσεις, ιδιαίτερα τη σύσταση υπαριθμών 6, που αναφέρεται στην εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οδηγία για τα ύδατα, την οδηγία πλαισίου για τα ύδατα, την ε, οδηγία για το πόσιμο ύδαρ και την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ. Να κλείσουμε το θέμα αυτό και θα κάνουμε ό,τι σας είπα πριν. Τώρα, συνεχίζουμε και περνάμε σε μια άλλη διαρευνητική επίσκεψη, η οποία έλαβε χώρα το Μάιο που μας πέρασε στην Αμόχωστο στην Κύπρο. Έχετε την έκθεση μπροστά σας. Ήμουν εγώ επικεφαλής της αποστολής. Και ήταν μια μεγάλη αποστολή, είναι αλήθεια, με πολλά μέλη και με τρεις εξοφίσιο. Ο αναφέρον ήρθε, μας συνάντησε, μας συνόδευσε σε επισκέψεις μας και είναι και εδώ παρόν σήμερα και τον ευχαριστώ πολύ, Λουίζο Αυξεντίου. Πολλά μπορεί να διαβάσει κανείς την έκθεση που προσπάθησα να ετοιμάσω βάσει γεγονότων, βάσει στοιχείων. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι πριν από 10 χρόνια η τότε Επιτροπή Αναφορών ήδη είχε πάει σε διαρευνητική επίσκεψη στην Αμόχωστο τότε. Τώρα, σήμερα, το μόνο που θα είχα να πω είναι ότι ο χρόνος πιέζει προκειμένου να βρεθεί μια συνολική λύση για αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι γεγονό ότι και από τις δύο πλευρές του νησιού οι άνθρωποι αρχίζουν να ξεχνάνε πώς είναι να ζουν μαζί και πώς είναι να μιλάνε ένα στη γλώσσα του άλλου. Αν λοιπόν θέλουμε μια συνολική λύση, τότε θα πρέπει να βιαστούμε, γιατί θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο περνάει ο καιρός. Ε, τα παιδιά μεγαλώνουν, οι μεγάλοι γερνάνε και ο κόσμος ξεχνάει πώς ήταν η κατάσταση πριν από το 1974, που περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη αποβιώσει, δεν τους έχουμε πια μαζί μας. Έχουμε ακόμα πρόσφυγες στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε η διερευνητική επίσκεψη ευαισθητοποιήθηκε ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα. Ε, ο συναισθηματισμός ήταν μεγάλος. Ε, πολλές φορές ήταν και άτυπες οι επαφές μας. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις, είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν λαμβάνει υπόψη της τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέμε εμείς. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να εντείνουμε λίγο τι συστάσει μα. Γι' αυτό και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη φορά. Την είπα το εκπρόσωπο για τι εξωτερικέ υποθέσει, το Συμβούλιο και όλε τι χώρε μέλη να υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το οποίο να ζητούν πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας εξαιτίας της ε, επίθεσής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τονίσουμε με αυτό το ψήφισμα ότι εφόσον δεν ε, συμμορφωθεί με τα ψηφίσματά μας 550, 94 κλπ για το 789, εμείς ομόφωνα συμφωνήσαμε κατά την επίσκεψη αυτή με τα όσα είδαμε και διαπιστώσαμε. Ξέρω ότι πολλοί θέλουν το λόγο και θα σας δώσω το λόγο. Λοιπόν, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες που έχουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Πεπαδράκη, που ήταν και παρόν στην αποστολή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά να σας ε, συγχαρώ και εσάς προσωπικά για την άψογη διοργάνωση της επίσκεψης στην Αμόχωστο. Για μένα, όπως γνωρίζετε, είχε και ένα πολύ ιδιαίτερα συνασηματικό ενδιαφέρον γιατί είμαι από την Αμόχωστο. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στις συστάσεις και νομίζω ότι οφείλουμε να το πράξουμε είναι ότι το θέμα της αμοχώς του είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα και θα πρέπει να το παραπέμψουμε για συζήτηση σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη στιγμή που η Τουρκία προσδοκεί να επαναχτίσει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να βγει από τα δικά της τα διέξοδα. Θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική ευκαιρία ούτως ώστε να ασκηθεί ουσιαστική πίεση για την παράδοση της πόλης της Αμχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, ξεχωρίζοντας από τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τη λύση του Κυπριακού. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και πρέπει να ασκηθεί πίεση ούτως ώστε να συζητηθεί ουσιαστικά το θέμα της Αμχώστου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς που ηγηθήκατε μια ευρεία, όπως έχετε πει, αντιπροσωπείας επίσκεψης στην Αμόχωστο και όλους βεβαίως τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν και που νομίζω ότι απέδειξαν με, την, με τις δηλώσεις τους αλλά και με τα όσα μας έχουν πει ότι κατανόησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο το τι τρέχει γύρω από το κυπριακό πρόβλημα, αλλά ειδικότερα για αυτή την εγκλωβισμένη κατεχόμενη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Λοίζον Αυξεντίου που χωρίς την ε, δική του κατάθεση αναφοράς πριν αρκετά χρόνια δεν θα, ήταν δυνατή αυτή η επανάληψη της επίσκεψης και βεβαίω όλους τους ε, Κύπριους που παρά τις δυσκολίες της ημέρας, γιατί ήταν εργάσιμη ημέρα και δεν μπορούσαν να είναι... Δεν, μπορούσαν, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους για να είναι εκεί. Παρόλα αυτά, εκατοντάδες άνθρωποι μας συνόδευσαν σε αυτή την επίσκεψη. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Είμαστε 44 χρόνια μετά την εισβολή και θα ήταν ψέμα να πούμε ότι μετά από αυτή την επίσκεψη δημιουργούνται πιθανότητε επιστροφής τη πόλη, άλλωστε δεν δημιουργήθηκαν τόσα πολλά χρόνια εγκύτερα προς το 74 προσπάθειες που ήταν ίσως και πιο εύκολο με ζωντανού πάρα πολλού από τους πρόσφυγες που προέρχονται από εκείνη την πόλη. Μπορεί όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Μα Κοινοβούλιο να κάνει κάτι παραπάνω. Πέραν από αυτά τα οποία έχει αναφέρει ο συνάδελφο ο κ. Παπαδάκη, νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαιτούν να επισκεφθούν την πόλη. Είχα ζητήσει παλαιότερα από τον κύριο Χάν, που είναι επίτροπος Διαβρύνσης και ασχολείται με θέματα Τουρκίας και Κύπρου συνακόλουθα, αφού η Κύπρος κομμάτι της μεγάλο κατέχεται, να επισκεφθεί την πόλη, ναι, να το ζητήσει. Να πούν όχι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδεικνύει κάθε ότι αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και δεν επιτρέπεται να κρατεί η Τουρκία του κατοίκου αυτή τη πόλη μακριά από τη γενέτειρα τους. Ιδιαίτερα μια πόλη που τα σπίτια έχουν εγκαταληφθεί, είναι μια πόλη ακατοίκητη, είναι ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεδομένου ότι ιδιαίτερα αυτή η πόλη συμπυκνώνει μεγάλο μέρο τη ευρωπαϊκή ιστορία. Μεγάλο μέρος τη ευρωπαϊκή ιστορίας. Το μαρτυρούν τα μνημεία της, οι εκκλησίε τη, τα τεμένη τη, τα τείχη τη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά από αυτή την επίσκεψη δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δοθεί εντύπωση στους ανθρώπους που κατάγονται από αυτή την πόλη κυρίω ότι κάναμε την επίσκεψη, κάναμε το καθήκον μας και εδώ τελειώνει. Πρέπει συνεχώς να εκπέμπεται το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιστοιχίζει την αγωνία αυτών των ανθρώπων και θα τους στηρίξει μέχρι την ημέρα της επιστροφής. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο λόγος είναι κύριο Μαυρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θα προσπαθήσω να μην προσθέσω, αλλά περισσότερο, να μην επαναλάβω, αλλά περισσότερο να προσθέσω σε όσα έχουν λεχθεί. Φυσικά οφείλουμε, και δεν είναι πλεονασμός, να συγχαρούμε εσάς ιδιαίτερα, αλλά και όλα τα μέλη που ταξίδεψαν στην Κύπρο και έχουν προσωπική αντίληψη της κατάστασης. Τι σημαίνει ένα έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υποξένη τουρκική παράνομη κατοχή. Προσωπικά, προερχόμενος από ένα άλλο μέρος της Βόρειας Κύπρου που είναι κατεχόμενη από την επαρχία της Κερίνιας, αισθάνομαι ιδιαίτερα και συμπάσχω βλέποντας και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτε μου, τα σπίτια μας να κατέχονται παράνομα. Όμως Αγαπητή κυρία Βίξτρομ, αυτό το θέμα ενώπιον μας θα προσπαθήσω να δώσω μια ευρύτερη διάσταση που είναι πολύ πέραν από την Κύπρο και έχει να κάνει και με τις επικείμενες ευρωεκλογές. Αυτός ο πολίτης, ο Ευρωπαίος εδώ από την Κύπρο, ο κύριος Αυξεντίου, με την ενέργεια του και την επιμονή του κατ' εμέ, φανερώνει την δύναμη αλλά και την αδυναμία του Ευρωπαίου πολίτη. Η δύναμη του είναι το γεγονός ότι με το βαροσότικο πείσμα του, εν και με τη βοήθεια πολλών άλλων, είμαστε εδώ και συζητάμε. Και ζητάει, τι ζητάει, το θεμελιακό δικαίωμα να απολαύσει το σπίτι που γεννήθηκε και του ανήκει. Αλλά ταυτοχρόνως, δυστυχώς, αυτή η υπόθεση φανερώνει και την αδυναμία των Ευρωπαίων πολιτών και δεν είναι τυχαίο που δυστυχώς όσοι πιστεύουμε και πιστεύουμε πραγματικά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την άποψη ότι η, θέση των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να αποκτήσει επιπλέον βαρύτητα ξεκινώντας φυσικά και από την αμόχωστο. Τελειώνω. Μια προσωπική ερώτηση προς εσάς. Διαβάζοντας προσεκτικά την έκθεση διαπιστώνουμε έχουμε μια φοβερή διαπίστωση ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να εφαρμόσει τα ψηφίσματα αλλά θέλει την αμόχωστο ως ένα διαπραγματευτικό ατού. Αγαπητή κυρία Σισίλια Γουίστρομ, πείτε μας επίσης τι νομίζετε, ποια είναι η πιθανή εξήγηση γιατί εκείνος ο Τούρκος διοικητής δεν προσέτρεξε στο κάλεσμά σας να σας επιτρέψει με την αποστολή να μπείτε στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Τώρα ο λόγος είναι για τον κύριο Χριστοφ... Χριστοφόρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά, αν και θα είναι πλεονασμό, εν τούτη όμω ε, οφείλω ευγνώμονε ευχαριστίε να επαναλάβω προ την Επιτροπή σα και εσά ιδιαίτερα προσωπικά που ηγηθήκατε αυτή τη αποστολή, μια αποστολή που μαζί με την ομάδα σα, σε όλων των συναδέλφων Ευρωβουλευτών, άγγιξε τι καρδιέ και τι ψυχέ όλων των Ελλήνων τη Κύπρου. Γιατί εκεί πήγατε για να δείτε η διεισόμαση, την ανίποτη τραγωδία που υφίσταται ο Κυπριακό Ελληνισμό εδώ και 44 χρόνια. Και ω Έλληνα Κύπριο, εκφράζοντα ολόκληρον τον Κυπριακό Ελληνισμό, πραγματικά οφείλω να υποκληθώ στην ε, ακατάπαυστη προσπάθεια που καταβάλλεται αισθανόμενοι και νιώθοντα, και αυτό είναι το σημαντικό και εσεί, ότι η πόλη τη Αμοχώστου δεν είναι μια ξένη πόλη, είναι μια ευρωπαϊκή πόλη και οι Αμοχωσκιανοί είναι Ευρωπαίοι πολίτε και το ίδιο αισθάνεστε και εσεί με όλου αυτού. Γι' αυτό σα ευχαριστώ, όπω ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην εξάρω την πρωτοβουλία του αγαπητού Λοίζου Αξεντίου, που στο πρόσωπό του αντανακλάται ο κάθε Έλληνα Κύπριο πρόσφυγα, ο οποίο απόλυσε την περιουσία του σήμερα το 2018 που μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, που μιλάμε για πρόσφυγες όπου γης, έχουμε 200.000 Ευρωπαίους πρόσφυγες που εκεί είναι τεράστια οφειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο για τους υπόλοιπους πρόσφυγες που καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μοριά ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της γης, αλλά για αυτούς τους 200.000 Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, Ευρωπαίους πρόσφυγες, δικαίως καθημερινά μας ρωτούν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας που είμαστε δικοί της πρόσφυγες και υφίστανται μάλιστα αυτήν την τραγωδία από μια χώρα που το διαπιστώσατε και μόνοι σας ότι είναι μια χώρα που έφερε την καταστροφή, την τραγωδία στον τόπο μας, την τραγωδία στην Αμόχωστο, μια πόλη την οποία κράτησαν ερυπωμένη εδώ και 44 χρόνια, απαγορεύοντας το βασικό και ανθρώπινο δικαίωμα των κατοίκων της να βρεθούν εκεί και να ζήσουν και να συνεχίσουν τη ζωή του. Ουσιαστικά το Ευρωκοινοβούλιο συνάντησε αυτόν τον σκληρό πρόσωπο τη κατοχή. Και δικαίω διαρωτάστε πώ είναι δυνατόν η Τουρκία να συνεχίζει να προπαγανδίζει ότι θέλει λύση του κυπριακού προβλήματο, όταν ένα ζήτημα όπω τη αμοχώ του, που θα μπορούσε μέσα σε μια μέρα να την παραδώσει στου νόημου κατοίκου τη και να απομακρυνθεί από αυτήν την τραγική κατάσταση, όχι μόνο δεν το πράττει, αλλά βιώσατε το σκληρό πρόσωπο τη κατοχή που δεν σα άφησαν να μπείτε σε ευρωπαϊκό έδαφο. Ποιο, ο Τούρκο διοικητή. Η Τουρκία εφαρμόζει τον νόμο τη βία των όπλων και τη δύναμη των όπλων. Το ζήσατε και το βιώσατε. Και ένα πολύ σημαντικό θέλω να πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο οφείλουν να κάνουν πολλά. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσει είτε σε χώρε μέλη είτε σε χώρε που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να έχουμε μια χώρα όπω την Τουρκία που παραβιάζει καθημερινά ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών. Αυτέ τι μέρε συνέλαβε ακόμα και αλλιευτικά σκάφη η Τουρκία καταδεικνύοντα ότι εκεί λειτουργεί ω πειρατή και τρομοκράτη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναλαμβάνει ευθύνη να επιβάλλει κυρώσει. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να στείλει το μήνυμα ότι σε αυτήν την Τουρκία που παραβιάζει κατάφορα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τη, που εφαρμόζει τον νόμο των όπλων και την πολιτική των κανονιοφόρων στη Μεσόγειο, δεν μπορούν να μην επιβάλλονται κυρώσει. Και να πω κάτι που ω Ευρωπαίων πολίτη με θίγει ιδιαίτερα. Οι Αμερικανοί για έναν Αμερικανό πολίτη επέβαλα στη σύμμαχο του Τουρκία που είναι σύμμαχο του για πολλά χρόνια επέβαλαν αυστηρέ κυρώσει σε βαθμό που ταρακούνησαν την Τουρκία. Ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρόσφατα συζητήσαμε ότι πρέπει να είναι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θέμα τη του και για τα άλλα ζητήματα οφείλουμε πραγματικά να αποδείξουμε ότι είμαστε ισχυροί και να μην χαριζόμαστε πλέον σε καμιά Τουρκία το ότι το ζήσατε εσεί τα γνωρίζετε καλύτερα πλέον από οποιοδήποτε άλλον και τα νιώθετε και σε εσά βασιζόμαστε γιατί πραγματικά Πιστεύω ακράδαντα ότι αισθάνεστε την αμόχωστον όπω την αισθάνεται ο καθένα από εμά πλέον και μπορείτε αυτή τη φωνή να τη μεταφέρετε ω Επιτροπή και μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε και ω Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και σίγουρα συμφωνώ αυτό το θέμα να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ πραγματικά για ό,τι κάνετε για όλου εμά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Θεοχάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε επισκεφτεί μαζί την Αμόχωστο αρκετές φορές και αρκετές φορές με τη συνοδεία του Λοΐζου Αυξεντίου, ο οποίο από το, από το 2004 πηγαίνω έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δικά του έξοδα, εγκαταλείποντας και την εργασία του και την οικογένειά του για να συντηρεί αυτό το ζήτημα. Ε, βεβαίως το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι μόνο πρόβλημα της αμοχώς του και δεν είναι μόνο πρόβλημα περιουσιών, είναι το πρόβλημα μιας ιστορίας χιλιάδων χρόνων που σβήνει και καταστρέφεται αυτό τον καιρό. Πρέπει να θυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι πριν από μερικά χρόνια οι Τούρκοι που κατέχουν την Αμοχωστό συνέλαβαν τέσσερις ευρωβουλευτές, την Ομιλούσα, τον Αρτούρ Ζασάτα, τον κύριο Βαλέσα, την νυν επίτροπο την κυρία Νεδέλτσεβα Γκάμπριελ, τον Λοΐζο Αυξεντίου και τον πρώην Ευρωβουλευτή Μάτσι, γιατί Κάναμε το αυτονόητο, να μπούμε μέσα στην πόλη της Αμοχώστου. Ακολούθησε ένα, μια written declaration από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το ποσοστό που εξελέγει ο Σούλτς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνη η γραπτή διακήρυξη μας έδωσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μην αφαιθεί να σβήσει από τις δέλτους της ε, Επιτροπής της petition, της petty committee, τα αναφορών, ναι, της Επιτροπής Αναφορών, σας ευχαριστώ, ε, το ζήτημα της αμοχώς του. Και θυμάστε στην πρώτη μας συνεδρίαση, ένα από τα σημεία αιχμής ήταν αν θα διαγράφαμε το ζήτημα της αμοχώς του. Θέλω να τονίσω το εξής η Τουρκία είναι ένα υβριδικό τρομοκρατικό κράτος. Τόσα χρόνια πολύ λίγοι άνθρωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καταλάβαιναν. Ο όγκος των συναλλαγών, βλέπετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι τεράστιος. Τώρα όμως που έχετε καταλάβει όλοι, εσείς το καταλάβατε πάρα πολύ νωρί, γιατί είχατε και φίλους Κύπριους που σας πήγαν και είδατε μέρη. Το ίδιο και πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές. Τώρα που το κατάλαβαν όλοι, οφείλουμε να επιβάλλουμε σκληρές κυρώσεις στην Τουρκία για να εφαρμόσει αυτά που προνοούνται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου του 1977 και του 1979 που προνοούν την άνευ όρων επιστροφή της πόλη, της πόλης της Αμοχώστου, αυτά που περιλαμβάνει η γραπτή διακήρυξη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και το χρέος μας προς την ηθική, το χρέος μας προς την ιστορία, το χρέος μας προς τον πολιτισμό η Κύπρος οφείλει να απελευθερωθεί και αυτή η ιστορία των δύο μερών που θα επανενωθούν θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι είναι μια ηλαροκομωδία. Ο λαός ζούσε διάσπαρτο σε όλα τα μέρη της Κύπρου, μειχτός, τεχνητά τον έχουν διαχωρίσει με τη βία των όπλων και δεν ήταν διασυνοριακή διαφορά του βορρά που ήταν κατεχόμενος από μουσουλμάνους και του νότου που ήταν κατεχόμενος από Έλληνες. Γι' αυτό το λόγο Ας κατανοήσουν επιτέλους όλοι το όνομα του, Κυπρια... του Κυπριακού. Θερμά ευχαριστώ τον φίλο Λοΐζο Αυξεντίου και σας βεβαίως για ό,τι κάνετε για την απελευθέρωση της Κύπρου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μα... Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ τον αναφέροντα, τον κύριο Λοΐζο Αυξεντίου, για τον αγώνα τον οποίο δίνει όχι βέβαια μόνο του, αλλά για λογαριασμό όλων των κατοίκων της αμοχώστου του και συνολικά για λογαριασμό του Κυπριακού λαού. Να πω επίσης ότι αποδεικνύεται η, πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή μας. Διότι πήραμε μια σωστή απόφαση σε επίπεδο συντονιστών, δηλαδή να γίνει αυτή η επίσκεψη, η οποία πραγματικά αναδεικνύει τα προβλήματα διότι άλλο είναι να κουβεντιάζουμε εδώ σε κλειστέ αίθουσε, άλλο είναι να έχουμε έστω και τον αναφέροντα και τους αναφέροντες να λένε τι συμβαίνει και άλλο πλέον να υπάρχει η εμπειρία προς τους ίδιους τους ευρωβουλευτές και φυσικά στους αναφέροντες και στους υπολείπους το τι εστί τουρκική κατοχή, τι σημαίνει να υπάρχει μια ολόκληρη πόλη φάντασμα που απαγορεύεται κανείς να εισέλθει, τι σημαίνει να υπάρχει στην Ευρώπη η μοναδική αυτή περίπτωση όπου υπάρχει μια ολόκληρη πόλη που την έχουν καταλάβει παράνομα τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει ενώ εκεί είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Φαίνεται λοιπόν πλέον η αναγκαιότητα για τη λήψη μέτρων. Διότι είδαμε να λαμβάνονται μέτρα και κυρώσεις έναντι τρίτων χωρών οι οποίες κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση παραβίασαν το διεθνές δίκαιο άλλων τρίτων χωρών. Εδώ λοιπόν έχουμε καραμπινά την περίπτωση ενός τρίτου κράτους της Τουρκίας που μάλιστα θέλει να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει και σχέση ε, σύνδεσης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει καταλάβει το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας Έχουμε, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι έχουν προκληθεί λόγω αυτού του γεγονότος, οι οποίοι δεν την χάνουν τη μέρημνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έπρεπε να την χάνουν, τουλάχιστον αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη μέρημνα όπως και άλλοι πρόσφυγες που έρχονται πλέον στην Ελλάδα ή στην Τουρκία ή και στην Κύπρο ακόμη. Και πλέον νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν τα λόγια διότι έχουμε την έκθεση, έχουμε αναλυτικά τι έχει συμβεί, έχετε φωτογραφίες, έχετε την απαγόρευση που υπήρξε από πλευράς των στρατευμάτων κατοχής των Τούρκων και πλέον αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθεί μια απόφαση για την συγκεκριμένη αναφορά και προτείνω κυρία Πρόεδρε να κάνουμε μια συζήτηση πλέον υπομορφή ε, ερωτήσεως προς το ε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί πολλά σημαντικά θέματα από αυτήν εδώ την Επιτροπή τα έχουμε οδηγήσει, όπως ξέρετε και με πρωτοβουλία δικιά σας, στην Ολομέλεια. Επομένως να φέρουμε το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχουμε επισημάνει μέσα στο δικό μας ψήφισμα την αναγκαιότητα πλέον λήψης συγκεκριμένων κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι οι ίδιοι οι αναφέροντες θα δικαιωθούν ή θα αρχίσει μια διαδικασία δικαίωση. Διότι το να μείνουμε απλά σε μια συζήτηση εδώ, η οποία βεβαίω είναι σημαντική και ένα ψήφισμα σημαντικό, μια έκθεση που θα μείνει μόνο σε επίπεδο Επιτροπή Αναφορών, νομίζω θα είναι μισό βήμα. Να πάμε παραπέρα, να το θέσουμε στην Ολομέλεια, να έχουμε προτάσει πολύ συγκεκριμένε και πρακτικέ, είτε να καλούμε Ευρωπαίου αξιωματούχου να επισκεφτούν την αμόχωστο και τον αρμόδιο επίτροπο τον κύριο Χάν όπως υπόθηκε αλλά και την κυρία Μογκερίνη και άλλους αξιωματούχους τον ίδιο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντιπροσωπεία διότι μόνο έτσι και συνοδευόμενοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διότι μόνο έτσι θα εκτεθεί διεθνώς η Τουρκία και θα αναγκαστεί να υποχωρήσει σε πιέσεις και δεύτερον να έχουμε και μέτρα και κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την πολιτική την παράνομη που ασκεί απέναντι στην Κύπρο ειδικότερα στην Αμόχωστο, στα κατεχόμενα και τώρα τελευταία με τις συλλήψεις τις παράνομες των αλλιευτικών των Κυπριακών. Μόνο έτσι πρακτικά μπορούμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά θα έχουμε κάνει μισό βήμα, σημαντικό, ότι πήγαμε, ότι είδαμε, ότι τα λέμε, αλλά να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, κυρία Πρόεδρε, το προτείνω σε εσά, η οποία θα μας προτείνετε τι μέτρα θα πάρουμε παρακάτω για να συνεχίσουμε αυτή την αναφορά και νομίζω ότι πηγαίνοντα το θέμα στην Ολομέλεια, ε, στο Στρασβούργο, θα είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα είναι το αναγκαίο επόμενο βήμα. Σας ευχαριστώ. Fine, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω εξαντλήσει τον κατάλογο μιλητών. Ξαφνικά έγινε πολύ Κύπρια και ελληνόφωνη η επιτροπή μας. Όμορφο αυτό. Τώρα βέβαια να ζητήσουμε και από τον αναφέροντα να πάρει το λόγο. Και μετά θα επανέλθω να σας πω γιατί η έκθεση έχει ως έχει και οι συστάσεις. Ο κύριος Αυξεντίου όμως τώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ποτέ δεν θα μάθω να προφέρω καλά το όνομά σας. the is yours and... Έχετε το λόγο και πριν αρχίσετε Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας συνοδεύσατε στο κατεχόμενο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αποστολής μας εκεί και στα Βαρόσια. Νομίζω ότι δεν θα ξεχάσει κανείς μας την επίσκεψη, το διάλογο που είχαμε έξω από το σπίτι σας. Εσείς είσαστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού ουσιαστικά μας προσκαλέσατε όλους και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσετε πραγματικά να μας προσκαλέσατε και για δείπνο σε αυτό το σπίτι. Βεβαίως, ένα πάρτι θα κάνουμε τότε, αν φτάσει αυτή η ευλογημένη μέρα. Κυρία Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της διερευνητικής αυτής επίσκεψης στην Αμόχωστο, αλλά και ολόκληρη την Επιτροπή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αιμονή σας από την αρχή, από το 2004 που υπέβαλα την αναφορά μου, 14 χρόνια τώρα. Έρχομαι και επανέρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Αναφορών, για να σας ενημερώνω για το τι συμβαίνει στην χώρα μου και στην πόλη μου. Όταν υποβάλαμε την αναφορά αυτή, θέλαμε πρώτα απ' όλα να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα έγκλημα το οποίο λαμβάνει η χώρα στην χώρα μας από το 1974, παραβίαση θεμελιωδών και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτή είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Έγινα πρόσφυγα στον Αύγουστο του 1974 και είμαι πρόσφυγα στα τελευταία 44 χρόνια. Παντρεύτηκα μία ε, πρόσφυγα και τώρα μεγαλώνω τους ε, γιους μου πρόσφυγες ε, και αυτοί, έναν από τους δύο τον γνωρίσατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση στην Κύπρο σήμερα και συνεχίζεται. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση βίας και διατηρείται με την χρήση βίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Κυρία Πρόεδρε, η αναφορά μας πηγαίνει ακόμα πιο πέρα. Στην πρώτη μου παρουσίαση εδώ σε αυτό το σώμα μίλησα για τη δήλωση Σούμαν και πιο συγκεκριμένα ζήτησα από τους ευρωβουλευτές να θυμηθούν μία φράση της δήλωσης αυτής, ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να φτιαχτεί μέσα σε μια μέρα ή με ένα μόνο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά με την ε, αλληλεγγύη που μας ενώνει. Αλληλεγγύη για τα θέματα τα οποία είναι κοινά μεταξύ μας. Και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε στην Αμόχωστο. Προσπαθούμε δηλαδή τους νόμιμους ιδιοκτήτες των σπιτιών που βρίσκονται στο εγκλωβισμένο μέρος να επιτρέψουν στα σπίτια τους. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να έχουμε σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους, αυτούς τους Τουρκοκύπριους που βρίσκονταν εκεί από την αρχή και εξακολουθούν να ζουν στην Αμόχωστο. Θέλουμε να υπάρξει αυτή η δημιουργία αλληλεγγύης μέσα στο νησί μας. Και εσείς κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε στην ε, πρώτη διαρευνητική επίσκεψη και είπατε ότι σιγά σιγά ξεχνάμε ε, το πώς ζούσαμε μαζί. Είναι αλήθεια. Αν επιστρέψουμε στα σπίτια μας θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε με τα αδέρφια μας τους Τουρκοκύπριους που είναι και αυτοί όσο Κύπροι είμαστε και εμείς κυρία Πρόεδρε. Είμαστε Ευρωπαίοι πρόσφυγες. Δεν ζούμε σε σκηνές πια, παρόλο που ζήσαμε για αρκετά χρόνια μετά το 1974 σε σκηνές. Ε, καταφέραμε να βρούμε σπίτια, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα σπίτια μας βρίσκονται σε αυτό το εγκλωβισμένο τμήμα, υποκατοχή. Και όχι μόνο υποκατοχή, αλλά και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, ότι δηλαδή βλέπουμε τα σπίτια μας κάθε μέρα να καταστρέφονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω που στις συστάσεις σας έχετε συμπεριλάβει και αυτό που πρότεινα όταν με ρωτήσατε τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Και είπα ότι όταν χώρες όπως η Τουρκία παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τότε η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που δεχτήκατε την σύστασή μου αυτή και προτείνατε κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ ευχαρίστως να φιλοξενήσω οποιοδήποτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει να έρθει στην Κύπρο, στην Αμόχωστο και να δει το σπίτι μου εκεί. Ευχαρίστως να σας πάω. Και ένα πράγμα θέλω να ε, σας ζητήσω. Όταν ε, ολοκληρώσετε το έργο σας εδώ στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, όταν επιστρέφετε στις χώρες σας και φτάνετε στην πόρτα του σπιτιού σας και είσαστε έτοιμοι να ξεκλειδώσετε την πόρτα σας, σας παρακαλώ να θυμηθείτε το δικό μου σπίτι το σπίτι μου έτσι όπως είναι σήμερα αυτή τη στιγμή σε μια εγκλωβισμένη ζώνη και κατεχόμενη. Θα ήθελα και εγώ να μπορώ να επιστρέφω στο σπίτι μου και να ανοίγω την πόρτα μου. Κάθε μέρα, εγώ όταν τελειώνω τη δουλειά μου, όπως κάνετε κι εσείς κάθε μέρα, γυρνάτε στο σπίτι σας και θα ήθελα και εγώ να μπορώ να κάνω το ίδιο. Είναι ένα δικαίωμα που έχω ως Ευρωπαίος πολίτης. Και είναι ένα δικαίωμα όμως που μου το αφαίρεσε μου το φέρει σε μένα, της οικογένεια μου, των ε, δικών μου, των συμπολιτών μου, η Τουρκία. Και αυτό είναι που πρέπει να διορθωθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβουμε ότι δεν θεωρούμε επιλογή το status quo. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την ημερομηνία, οπότε θα μπορέσετε και εσείς να επιστρέψετε μαζί με τους υπολείπους στο σπίτι σας. Εδώ είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να σας καλέσω να μας πείτε τις σκέψεις σας επί της έκθεσης. Έχετε διαβάσει πολλές εκθέσεις για διαρευνητικές επισκέψεις και για το ίδιο θέμα. Αλλά βλέπετε ότι ο μορφότυπος της έκθεσης αυτής διαφέρει από τις προηγούμενες, καθώς έχει μόνο μία σύσταση. Και θα ήθελα να αντιδράσετε για τη σύσταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. η επιστροφή της φραγισμένη περιοχή των Βερουσίων στην Αμόχωστό στου νόμιμου κατοίκους αναμένεται να είναι ένα από τα κύρια σημεία των διαπραγματεύσεων για να υπάρχει μια βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαπραγματεύσεις αυτές, αν ξαναξεκινήσουν, θα είναι υπό την ηγεσία της Κύπρου και την καθοδήγησή της. Ε, εμείς ε, θέλουμε να πούμε ότι μια επίλυση που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ε, γιατών της Κύπρου θα αποτελεί το πιο μέσο τρόπο να επιληθεί το πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την επιστροφή των βερουσίων στους νόμιμους ιδιοκτήτες του. Σύμφωνα με την πάγια δέσμευση ε, για την επίλυση του Κυπριακού, η Κομισιόν είναι έτοιμη να υποστηρίξει πολιτικά καθώς και τεχνικά τις προσπάθειες των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αλλά και των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρξει μία πλήρης επίλυση του Κυπριακού. Ιδίω η Κομισιόν είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα σχετικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνονται από τις δύο κοινότητες ε, και σε ό,τι αφορά τα βαρόσια. Επίσης, να δράξω την ευκαιρία να σχολιάσω ένα σημείο στην έκθεση για να επικαιροποιήσω την κατάσταση σε σχέση με τα σημεία διέλευσης. Ε, ολοκληρώνονται τα έργα και τα κύρια ζητήματα τώρα ε, υπάρχουν στην ελληνοκυπριακή πεδρά. Το ένα αναφορά ένα σημείο διέλευση στη Δερίνια. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Κομισιόν ε, επανειλημμένα έχει υπογραμμίσει μεταξύ άλλων και στην η έκθεση 2018 για την Τουρκία ότι η Τουρκία αναμένεται να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και πλήρη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι βουλευτές ε, θα ήθελαν να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κύριος Σόλτες ε, ήταν και στην αντιπροσωπεία, συμμετείχε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο. Είχαμε ενεργή συμμετοχή άλλων συναδέλφων ε, από την Κύπρο και γι' αυτό εγώ δεν ε, ήθελα να παρέμβω. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πολύ συγκεκριμένο, αλλά ελπίζω ότι η δική μας επίσκεψη δεν ήταν, να μην είναι η τελευταία δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελπίζω να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στι ε, σχετικέ αρχέ, στι αρμόδιε αρχέ, όχι μόνο εντό αλλά και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο για να υποστηρίξουμε, αλλά για να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιστραφούν τα σπίτια και η γη στους αναφέροντες. Γιατί αν θέλουμε να περασπίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και τα πρότυπα, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, δράσεις μας για να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω τον κύριο Μαυρίδη. Κύριε Μαυρίδη, θέλετε να συμπληρώσετε, παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλούμε. Just 30 seconds. Um... δευτερόλεπτα. Θα ήθελα μια απάντηση για την ερώτησή μου από εσά. Αλλά επίση να πω ότι δεν μπορώ να το αφήσω αυτό χωρίς κανένα σχόλιο. Θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου, γιατί η έμφαση δίνεται από την Κομισιόν στην ε, τελική επίλυση του Κυπριακού. Είναι και δική μα επιθυμία αυτό. Αλλά αυτά που συζητάμε σήμερα δεν είναι η επίλυση του Κυπριακού. Συζητάμε συγκεκριμένα την εφαρμογή δύο ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ό,τι αφορά την αμόχωστο και ειδικά τα βαρόσια και πώς θα πιέσουμε για το θέμα αυτό να επιστραφεί η αμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους και διοκτήτε τη, όπως είναι ο κύριο Αυξεντίου. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να λάβετε θέση και όχι γενικά να το γενικοποιήσετε το θέμα και να αναφέρεστε μόνο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ηγετών της Κύπρου. I could have... Κοιτάξτε, θα μπορούσα να έχω επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο διάρθρωσης της έκθεσης. Εγώ διάλεξα αυτόν και ηλεκτρονικά έχετε λάβει τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες και σήμερα έχετε λάβει και την έντυπη μορφή στους φακέλους σας. Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε από μένα και έχει σταλεί σε όλα τα τακτικά μέλη της αντιπροσωπείας και με ικανοποίηση σας ενημερώνω ότι έχουμε φτάσει σε πλήρη συνένεση, σε συμφωνία με όλες τις ομάδες για το περιεχόμενο δηλαδή δεν θα παρουσιαστεί τροπολογία για τον τελευταίο παράγραφο. Βλέπετε ότι έχω προτείνει μόνο μία σύσταση. Επομένως, είναι ε, από πολιτική σκοπιά κάτι που πηγαίνει πολύ μακριά δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες ούτε αναφέρεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πολλά θα μπορούσαμε να έχουμε προσθέσει για το γεγονότα, θα μπορούσα να αναφερθώ στο πώ στάθηκα στο να στέκομαι μπροστά στην πύλη και να έχω τον Τούρκο διοικητή να προχωράει εναντίον μου. Ήμουν εκεί μόνη μου και όταν με είδε έστρεψε και έφυγε από την άλλη. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και να πυροδοτήσω αυτή τη, σύραξη, τη σύγκρουση, αλλά διάλεξα ένα διαφορετικό τρόπο και με υποστήριξαν όλα τα κόμματα. Τώρα, είχαμε εδώ μία συζήτηση και θα πρέπει να βρούμε κοινή θέση για να προωθήσουμε τον κοινό στόχο με τον οποίο συμφωνούμε όλοι, δηλαδή την επιστροφή των βεροσίων στους νόμιμους κατοίκους τους 44 χρόνια, σχεδόν 45 μετά την τουρκική εισβολή. Σε αυτό σκοπεύουμε. Προσπαθήσαμε και κάθε διεθνής παίκτη. Ε, έχει καταβάλει απόπειρες όλες οι τρεις προσπάθειες 2005, 2006, 2010 από τις Προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτύχει. Επίσης, ε, το Μάιο του 2014 είχαμε και το master plan ε, του κυρίου Μπάιντεν για την αμόχωστο και περιλαμβανόταν ε, εκεί η επιστροφή των βεροσίων υπό τη δίκηση του ΕΕ με ανταλλαγή άλλων στοιχείων. Όλα αυτά έχουν αποτύχει μέχρι τώρα. Η πρόταση που ε, έχει υποβληθεί από τους ελληνικυπρίους ηγέτες για την επιστροφή των βεροσίων δεν έχει επιτυχίας. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να κλιμακώσουμε την πίεση και ε, στην διάσκεψη των Προέδρων να πάμε το θέμα αυτό, να τους πιέσουμε, να τους κάνουμε να κάνουν το επόμενο βήμα και γι' αυτό βλέπετε αυτή τη σύσταση σήμερα. Γιατί αν το θέτουμε αυτό, αν το θέσουμε αυτό στο Συμβούλιο και χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε εδώ και εκπρόσωπο της Αυστρικής Προεδρίας του Συμβουλίου, θα σας έρθει αυτό, θα πάει στην διάσκεψη των Προέδρων και θα στη συνέχεια θα το προωθήσουμε. Αυτά έχω να πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπρόσθετα, τροπολογίες για τη σύσταση, που όπως σας είπα είναι μία. Προθεσμία είναι Παρασκευή αυτή την εβδομάδα στις 3 το απόγευμα και η ψηφορία στην Επιτροπή θα λάβει χώρα στις 21 Νοεμβρίου. Αυτά νομίζω. Τώρα όλοι θέλετε να δευτερολογήσετε. Ξέρετε, θα φύγουν οι διερμηνείς. Την Εντάξει, πολύ γρήγορα τότε. Λέω να χαιρετήσουμε την παρουσία στην αίθουσα του Αντιδημάρχου Αμοχώστου του Χρυσανθού Ζανέτου και του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοχώστου που είναι στην αίθουσα. Εάν νομίζετε σωστό, εγώ το θεωρώ να πούν δύο λόγια. Εάν όχι, μπορείτε να συνεχίσετε όπως έχετε καθορίσει. Ευχαριστώ. Ε, πολύ γρήγορα, να αφήσουμε και ανοιχτή την οψιόν το ενδεχόμενο να φέρουμε το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συζήτηση και ψήφισμα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχουμε διαδικασίες εδώ στο Κοινοβούλιο, δηλαδή ψηφίζουμε στην Επιτροπή και αν είναι απαραίτητο καταρτίζουμε ψήφισμα. Χρειάζεται όμως οι συντονιστές να λάβουν σχετική απόφαση. Σήμερα λοιπόν κάναμε ένα βήμα και σας είπα πώς θα προχωρήσουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι Καλή επιστροφή στην πιο όμορφη γωνιά της Ευρώπης. Και το λέω αυτό κοιτώντας τον αρκετά γκρίζο ουρανό των Βρυξελών. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τους χαιρετισμού μας και πριν ε, κλείσουμε το θέμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία που έκαναν εξαιρετική δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Όπως και σε όλα θέματα άλλωστε. Μερικές φορές ξεχνώ να σα να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ όμως ολόκαρδα για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ για την προετοιμασία της διερευνητική επίσκεψης και την κατάρτιση του προγράμματος. Είναι εδώ αναπληρωτή Δήμαρχο τη Αμοχώ του. Έχουμε πολλού προσκεκλημένου από την ε, αμόχωστο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε το λόγο, πρέπει να προχωρήσουμε. Και εφόσον ε, οι Κύπροι ευρωβουλευτές ε, μίλησαν τόσο πολύ, ε, σας έφαγαν όλο το χρόνο. Όχι οι Έλληνες, οι Κύπροι. Εν πάση σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ας προχωρήσουμε γρήγορα στην ετήσια έκθεση που είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είμαι συγγήτρια και πάντα πολύ ευχαρίστω συζητώ το θέμα αυτό μαζί σα. Το πιο σημαντικό πράγμα που κάναμε πέρσι ήταν ο διάλογος με τους αναφέροντές μας και εδώ και κατά τις διαρευνητικές μας επισκέψεις και μέσω ε, ε, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κλπ. Ε, το επίκεντρο συνήθως ήταν τα περιβαλλοντικά θέματα, ε, τα απόβλητα, η διαχείριση του νερού και άλλα. Άλλα θέματα ήταν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα του παιδιού, ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, καθώς και κοινωνικές υποθέσεις όπως είναι οι συνθήκες εργασίας σε διάφορα κράτη-μέλη. Ένας από τους στόχους μας ε, ήταν ε, να συνεργαζόμαστε στενά με τις νομοθετικές επιτροπές ε, και νομίζω ότι η συνεργασία αυτή είναι καλύτερη κάθε χρόνο. Χαίρομαι που οργανώσαμε διάφορες ακροάσεις σε συνεργασία με άλλες επιτροπές και είχαμε πολύ επικοδομητική συνεργασία. Το δίκτυο PETINET ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο και θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Ελπίζω και πιστεύω ότι η αυξημένη συνεργασία θα αποτελέσει καλή βάση για την Επιτροπή μας και κατά την επόμενη θητεία. Ποιος ξέρει αν θα είμαστε εδώ και τι ρόλο θα παίζουμε. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ο φυσικό εταίρο μα στα θέματα αυτά, για την πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια του έτου. Σχεδόν το 1 τρίτο των αναφορών που λάβαμε είχε, ε, διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, λαμβάνουμε ε, απαντήσεις όλο και πιο σύντομα και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας για την εντήσια έκθεση και όπως πάντα να συνεχίσω τη συνεργασία μαζί σας. Στόχος μας είναι να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε την ε, έκθεση φέτος ε, τον Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Θα κλείσω εδώ και θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές, στους κοιόδης συζητητές. Αν θέλει να συνομιλήσει μαζί μου οποιοδήποτε από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία, θα είμαι ελεύθερη σε λίγα λεπτά. Θα έρθω έξω και θα μιλήσω μαζί σα. Λοιπόν, ο κύριο Σόλτε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να συναντήσετε τι Κυπριακέ Αντιπροσωπείε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι πολύ σύντομο. Γενικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ για την εκπόνηση του εγγράφου αυτού. Σε κάποια σημεία όμως έχω κάποιες επικρίσεις. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πραγματικό πρόβλημα εδώ. Ναι, πράγματι, κάθε χρόνο η Επιτροπή Αναφορών ε, λαμβάνει όλο και λιγότερες αναφορές δεν είμαι όμως πεπισμένος ότι ο λόγος γι' αυτό είναι η καλύτερη κατάσταση στις χώρες της Ευρώπης. Φοβάμαι ότι ο λόγος είναι άλλος. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ε, λιγότερες ε, παρατυπίες ε, ή κακή εφαρμογή των νόμων, ιδιαίτερα στον τομέα των θεμελιωδών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είμαι βέβαιος ε, αν οι πολίτες γνωρίζουν ότι οι αναφορές είναι ένα ε, εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους σε περίπτωση ε, παραβιάσεων στη χώρα τους ή μήπως δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν βλέπουν να έχει νόημα το να υποβάλουν αναφορές. Πιστεύω ότι σκοπός των αναφορών είναι να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους πολίτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο ανάμεσα στη χώρα του και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι μπορούν να μα ενημερώσουν για το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του στου διάφορου τομεί που αναφέρατε. Κατά καιρούς όμως έχω την εντύπωση ότι ο αναφέρον πρέπει να περιμένει πολύ για να λάβει απάντηση από εμάς ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό οδηγεί σε απογοήτευση και προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με την χρησιμότητα ολόκληρου του θεσμικού οργάνου. Οι πολίτες πρέπει να πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η Επιτροπή Αναφορών. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο σαφής και πιο ακριβής στις απαντήσεις που δίνει. και όχι να ε, κρίνει μη παραδεκτές τις περισσότερες αναφορές ε, εξ αρχής. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά το παραδεκτό. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια δεν θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις λόγω της πολιτικής πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ. Πάντως, όπως και να έχει, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ε, να σας συγχαρώ για την έκθεση που έχετε υποβάλει ε, νομίζω ότι πιάνετε τα κυριότερα ζητήματα που μας απασχόλησαν την προηγούμενη χρονιά. Βεβαίως θα υποβάλουμε και εμείς ορισμένες τροπολογίες για να βελτιωθεί, αλλά στις γενικές γραμμές θα έλεγα ότι τα συμπεράσματα είναι σημαντικά. Να επισημάνω τρία-τέσσερα μικρά θέματα. Πρώτον, θεωρώ πολύ σημαντική τη συνεργασία της Επιτροπής Αναφορών με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Νομίζω ότι διαμορφώνεται έτσι μια συνεργασία ουσιαστική, ούτω ώστε να καλυφθούν όλες οι πλευρές προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσα από τις εργασίες της δικές μας, είτε σε επίπεδο ε, κακοδιοίκηση αν υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Δεύτερον, θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι πήραμε ε, τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για το ζήτημα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με συζήτηση που κάναμε εδώ με τον κύριο Τίμερμανς με το τι πρέπει να αλλάξει διότι είμαστε σε μια εποχή όπου οι πολίτες πρέπει να έχουν το λόγο πρέπει αυτό το σημαντικό μέτρο που λέγεται Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία πραγματικά να αποκτήσει σάρκα και οστά, να γίνει πολύ πιο εύκολη η δυνατότητα εφαρμογής της και να αισθάνονται οι πολίτες ότι συμμετέχουν άμεσα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι αυτή η Επιτροπή ασχολήθηκε πάρα πολύ με το ζήτημα του Brexit. Και αν το δει κανεί, θα δει πραγματικά ότι σε ένα κορυφαίο πολιτικό θέμα, όπου είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της Βρετανίας έρχεται μέσα σε αυτή την Επιτροπή, τη δικιά μας Επιτροπή, ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών της Βρετανίας αλλά και άλλων πολιτών που θέτουν ζητήματα ενώ επί της ουσίας το θέμα είναι θα έλεγα διακρατικό. Αν θα μείνει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγει. Και όμως μέσα από την Επιτροπή μας νομίζω ότι δώσαμε την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες και στους Βρετανούς πολίτες οι οποίοι πολλοί από αυτούς διαφωνούσαν να εκφράσουν την άποψή τους. Πολλοί πολίτες των άλλων κρατών μελών να εκφράσουν την ανησυχία τους. Θα έχουν δικαιώματα αύριο στη Βρετανία. Τι θα γίνει σε περίπτωση ενός Brexit αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, εγώ τουλάχιστον μελετώντας και γράφοντας για την Επιτροπή Αναφορών από το 1992-93, δεν είχα δει ότι ενδεχόμενα θα έχουμε μια τέτοια διάσταση. Δηλαδή οι πολίτες αυτοτελώς σε αυτή την Επιτροπή σε μεγάλο βαθμό είτε να συμφωνούν είτε και να διαφωνούν με πολιτικές των κρατών ε, μελών σε σχέση με την ένταξή τους. Και το άλλο σημείο, και με αυτό κλείνω, είναι τα θέματα που συζητήσαμε γύρω από την παιδική πρόνοια. Τα θέματα αυτά μας απασχόλησαν, ήταν πολύ σημαντικά, όπως η ειδικότερη μορφή που απέκτησε αυτό το θέμα και το συζητήσαμε στην Ισπανία με τη διερεύνηση των αναφορών για εικαζόμενες αλλά σε μεγάλο βαθμό απεδείχθη κλοπές νεογέννητων βρεφών από νοσοκομεία κατά τη διάρκεια μετά τη δικτατορία κατά τη διάρκεια και μετά τη δικτατορία του Φράγκο. Ένα σοβαρό θέμα που απασχολούσε και απασχόλησε την κοινωνία τη Ισπανία. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε καλύψει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Τα κλασικά θέματα βεβαίω, τα δικαιώματα των πολιτών, περιβαλλοντική προστασία, ελεύθερη κυκλοφορία, αναγνώριση ε, προσόντων, αλλά και αυτές τις εξειδικευμένες περιπτώσεις που νομίζω ότι δίνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φόρτη μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς ε, ακούγοντας την προηγούμενα σημεία συνειδητοποίησα και πάλι τη σημασία της Επιτροπής σας και του έργου των μελών σας προκειμένου να δημιουργήσετε γέφυρες μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργανών και των πολιτών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά και συμπληρώνει άλλα είδη πρωτοβουλειών προς τους πολίτες. Όμως η δουλειά που κάνατε εσείς είναι πάρα πολύ θετική. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, Πρόεδρε. Τα προκαταρκτικά μας σχόλια είναι τα εξής. Καλωσορίζουμε όλα τα σημεία που έχετε θίξει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αφορούν ε, πρακτικές στοιχές, τη συνεργασία μεταξύ της ε, Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και μπορώ να πω και να επιβεβαιώσω ότι κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά από κοινού. Φυσικά με τις προθεσμίες έχουμε ένα θέμα. Τώρα για την ποιότητα των απαντήσεων Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και δεσμευόμαστε και ο πρώτος σίγουρα θα επιβεβαιώσει ότι προσπαθούμε να παρέχουμε καλύτερες απαντήσεις. Σε ό,τι φορά τα θέματα, σίγουρα και εμείς έχουμε ανησυχίε όπως το περιβάλλον, οι αναπηρίες, η ευημερία των ζώων, η προστασία των παιδιών, το Brexit. Και υπάρχουν και άλλα, τα οποία ξέρετε ότι εξακολουθούμε να είμαστε στη συζήτηση με το Κοινοβούλιο Παραδείγματο Χάρη το θέμα τη Χάρτα ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη ερμηνεία τη Χάρτα. Αλλά φυσικά το αφήνω αυτό για να συζητηθεί στην Ολομέλεια, όπω και διαδικασίε επί παραβάση. Ξέρετε ότι καθημερινά προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία διασφαλίζοντα βέβαια ότι εφαρμόζεται σωστά το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά δίνοντα και μια δεύτερη ευκαιρία σε όσου ήχου δεν έχουν τα μέσα να εφαρμόσουν άμεσα τον νόμο. Έτσι λοιπόν υπάρχει διάλογο με τα κράτη-μέλη και υπάρχει και δυνατότητα τα κράτη-μέλη που πιστεύομαστε ότι δεν συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να προετοιμάσουν τα επιχειρηματά τους και να τα παρουσιάσουν. Έχουμε λοιπόν αυτό το διάλογο που λαμβάνει χώρα και θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο που να διατηρεί το δικαίωμα της υπεράσπισης κατά κάποιο τρόπο. Εκτιμούμε λοιπόν ε, το έργο που κάνετε. σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις αναφορές, αλλά και τις διερευνητικές επισκέψεις και τις ακροάσεις που επιτρέπουν να ακουστούν όλες οι φωνές στην Ήπειρο αυτή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια ακόμη καλύτερη συνεργασία το επόμενο έτος. Αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτό. Προθεσμία καταθέση τροπολογιών θα είναι στις 27 του μήνα, στις 3 το απόγευμα θα ψηφίσουμε στις 21 Νοεμβρίου και σας εύχομαι καλό βράδυ.